Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα πρότεινα να ξεκινήσουμε. Καταρχήν να σας ενημερώσω ότι έχουμε διερμηνία σε όλες τις επίσημες γλώσσες, με εξαίρεση τα Ιρλανδικά, Γοεδελικά, Κελτικά. Και φυσικά να μεταδίδεται, στο, μεταδίδεται ζωντανά στο διαδικτύο αυτή η δημοσία ακρόαση και όλες οι ομιλίες θα μαγνητοσκοπηθούν. Με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να σας καλωσορίσω καπιτά μέλη και καλεσμένοι σε αυτή την διακοινοβουλευτική διάσκεψη που συνδιοργανώνεται από τις Επιτροπές Αναφορών και Νομικών Υποθέσεων με συμμετοχή της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας. Θα είναι μια καλή ευκαιρία να ανταλλάξουμε τις απόψεις και τις βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου γιατί νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η μεταφορά ε, και η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου δεν είναι τεχνικό θέμα, είναι κέρια σημεία και νευραλικά για την ε, δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ξέρουμε ότι αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως κρίση στο κράτος δικαίου ε, μείωση τη εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στη δυνατότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τι υποσχέσει που δίδει. Οπότε η αποτελεσματική εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, του ενωσιακού δικαίου, έχει κρίσιμη σημασία για την αξιοπιστία και την ε, νομοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το ενωσιακό δίκαιο μπορεί να αποφέρει αυτά αποτελέσματα στους ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις επιχειρήσει μόνο όταν εφαρμόζεται σωστά στην πράξη όταν δεν εφαρμόζεται σωστά ή εμπρόθεσμα η ενωσιακή νομοθεσία, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στερούνται των πλονεκτημάτων της. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντική η σημερινή αυτή διάσκεψη, γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε τη δέσμευσή μας και να εξασφαλίσουμε οι στόχοι πολιτικής και ε, η ενωσιακή νομοθεσία και τα αποτελέσματά της δεν ε, θα μειώνονται στη διαδικασία ε, μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, στην εθνική Ενωμητάξη. Γιατί τα κράτη-μέλη δεν υποχρεούνται μόνο να μεταφέρουν στην Ενωμητάξη του στο ενωσιακό δίκαιο, αλλά να εξασφαλίζουν και την εφαρμογή, γιατί οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουν ε, αλλάξει από τη σύνθηκε της Λισαβόνας και η κοινοβουλευτική συμμετοχή είναι πιο έντονη στη διαμόρφωση των πολιτικών και στην ε, νομοπαρασκευιστική διαδικασία υπάρχει καλύτερο διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπάρχει μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με τις νομοθετικέ προτάσεις, δυνάμει τη αρχής τη επικουρικότητας. Γι' αυτό και η συμμετοχή των κοινοβουλίων είναι πολύ πιο σημαντική, γιατί αυξάνεται η νομοποίηση των ε, κοινοτικών δράσεων χάρη στην κοινοβουλευτική συμμετοχή. Τα εθνικά βέβαια κοινοβούλια δεν είναι τα μόνα που συμμετέχουν στη διαδικασία εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Ε, και τοπική περιφερειακή φορείς, αλλά και τα εθνικά δικαστήρια εφαρμόζουν ε, επιτόπου το ενωσιακό δίκαιο και έχουν υποχρέωση να εξασφαλίσουν ε, και οι συνομοθέτες σαφή νομοπαρασκευαστική διαδικασία που θα στηρίζεται σε επιστήρια. Και μόνο μια τέτοια σωστή νομοθεσία μπορεί να εφαρμοστεί και πιο εύκολα και αποτελεσματικά και να αντιληφθούν οι πολίτε τα δικαιώματα και τι υποχρεώσει του και τα κράτη-μέλη, αρμόδιοι φορεί να μπορούν να εφαρμόζουν αυτό το νοσιακό δίκαιο. Ελπίζω λοιπόν να είναι ενδιαφέρουσα αυτή η μέρα για την ανταλλαγή απόψεων και θα δώσω αμέσω το λόγο στον συνάδελφο Πολ Σάκη, που είναι αντιπρόεδρο τη Επιτροπή ε, Αναφορών, τη Επιτροπή ΠΕΤΗ, όπω λέμε. Αλλά θα μα ε, συστηθείτε εσεί Ευχαριστώ. Ε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμοι καλεσμένοι, αξιότιμα μέλη της διάσκεψης. Με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους εκ μέρους Επιτροπής Αναφορών σε αυτή την διοργάνωση. Καλωσορίζω όλους συμμετέχοντες σε αυτή τη διακοινοβουλευτική συνεδρίαση που συνδιοργανώνει η Επιτροπή Αναφορών με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διαμεσολαβητών. Στη διάρκεια της συνεδρίασης θα μιλήσουμε για την εφαρμογή και εκτέλεση του κοινοτικού δικαίου και ε, να δούμε κατά πόσο ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών που έχουν εκφράσει ανησυχίες για την κακή εφαρμογή ή παραβίαση του ενωσιακού δικαίου, κυρίως υποβάλλοντας μεγάλο αριθμό αναφορών για τα θέματα αυτά, παραβίαση κακής εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου. Και μάλιστα ε, δύο μελέτες που θα παρουσιαστούν σήμερα θα σχολιάσουν κάποια τμήματα της ε, ενωσιακής νομοθεσίας που αποτέλεσαν το αντικείμενο πολυάριθμων αναφορών στην Επιτροπή Αναφορών. Καταρχήν, η οδηγία του 2014 για την αξιολόγηση των επιπτώσεων κάποιων ιδιωτικών και δημοσίων σχεδίων για το περιβάλλον και επίσης ένας κανονισμός του 2004 2014 μάλλον, για τα δικαιώματα των επιβατών των αερομεταφορών. Το περιβάλλον και τα δικαιώματα των καταναλωτών είναι δύο τομείς για τους οποίους οι πολίτες πιστεύουν ότι θα, το ενωσιακό δίκαιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί καλύτερα σε εθνικό επίπεδο. Και μάλιστα γι' αυτό έχουμε και παρουσία εθνικών βουλευτών παρουσία της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας και ένα εξαιρετικό επιτελείο εμπειρογνωμόνων και θα συζητήσουμε όλα αυτά τα σημαντικά θέματα σήμερα σε αυτή την ακρόαση. Σας εύχομαι λοιπόν μια καρποφόρα συζήτηση και επικοδομητική και δώσω το λόγο στην κυρία Σελίν Κάουερ που είναι γενική γραμματέας, ε, Γενική Γραμματέα Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα μας μιλήσει για τη σημερινή ακρόαση. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ και μπορώ να σας παρουσιάσω ε, κάποια εισαγωγικά λόγια για την ε, σημερινή ακρόαση στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής ε, νομοθεσίας. Όπως τόνισε και ο πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, η αποτελεσματική εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου είναι απολύτως αναγκαία έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν στο μέγιστο ε, τα ωφέλη της ευρωπαϊκής πολιτικής. Στόχος είναι λοιπόν να απολαμβάνουν τα δικαιώματα που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αλλά και να έχουν την δυνατότητα γρήγορα και αποτελεσματικά να χρησιμοποιούν ε, τα ε, προβλεπόμενα ένδικα μέσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί την ε, διαδικασία επιπαραβάση προ όφελο όλων μα, έτσι ώστε να διασφαλίσει πώ ε, το ενωσιακό δίκαιο εφαρμόζεται ε, σωστά. Θα ήθελα να σα πω δύο λόγια σχετικά με αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πριν από λίγα χρόνια, εγκρίθηκε μια ανακοίνωση για μια περισσότερο στοχευμένη στρατηγική προσέγγιση σχετικά με την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου είχε τίτλο «Καλύτερα αποτελέσματα μέσω καλύτερης εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου». Ε, η αρχή αυτή έχει δύο άξονες. Πρώτον, καλή συνεργασία με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να εξασφαλίσει την σωστή εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, διότι η πρόληψη είναι φυσικά καλύτερη από την θεραπεία. Και η πρόληψη μπορεί να γίνει ακριβώς με αυτή τη στενή συνεργασία με τις ε, Εθνικές Αρχές και τα Εθνικά Κοινοβούλια για την ε, μεταφορά του ενωσιακού δικαίου στην Εθνική Νομοθεσία. Η, η ανακοίνωση αυτή έχει στόχο να παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για τη μεταφορά ε, του ενωσιακού δικαίου από τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά επίσης να παρέχει την δυνατότητα αντιμετώπισης ε, καταγγελιών σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται σωστά μια οδηγία. Αντί λοιπόν να τρέξουμε στο δικαστήριο, προσπαθούμε να εισέλθουμε σε ένα διάλογο με τα κράτη-μέλη για να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις και να γεφυρώσουμε τα κενά. Έπειτα, η πολιτική εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει να κάνει με την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και την ε, απαλυφή των εμποδίων μέσω του διαλόγου καταρχάς. Υπάρχουν τέσσερις προτεραιότητες για να γίνει παρέμβαση από την Κομισιόν. Πρώτον, οι περιπτώσεις όπου η μεταφορά δεν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει με τον κατάλληλο τρόπο στο εθνικό δίκαιο. Δεύτερον, περιπτώσεις όπου τα κράτη-μέλη δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Τρίτον, υποθέσεις όπου διακυβεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Και τέλος, υποθέσεις όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα. Αυτές λοιπόν είναι οι τέσσερις προτεραιότητες που έχουμε θέσει και αναγνωρίζουμε βέβαια πλήρως ότι τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις αυτό γιατί η προσέγγιση δεν είναι και η πιο εύκολη. Θεωρούμε όμως ότι η συνεργασία είναι ουσιώδης και γι' αυτό υπάρχει και ο ρόλος της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας ως πρώτο σημείο επαφής έτσι ώστε να ε, γίνονται γνωστά τα προβλήματα των πολιτών. Οι έρευνες οδηγούν σε έβρεση περιπτώσεων που όντως έχει παραβιαστεί το ενωσιακό δίκαιο. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε πως η συνεργασία αυτή καθιστά μια πραγματική εταιρική σχέση. Έχουμε ήδη διοργανώσει τις πρώτες ε, συνεδρίες συνεργασίες ανάμεσα στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε πνοή σε αυτήν την συνεργασία. Ελπίζουμε σύντομα να καταφέρουμε να διοργανώσουμε και δεύτερη τέτοια ε, ομάδα εργασίας. Επίσης, το Σεπτέμβριο το Ελεκτικό Συνέδριο δημοσίευσε μία σύνοψη της ε, κατάστασης ε, μεταφοράς του νοσιακού δικαίου στην εθνική νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Νομίζω πως ε, στην έκθεση αυτή αναγνωρίστηκαν οι προσπάθειες της Κομισιόν για την βελτίωση της ε, κατάστασης σχετικά με την ε, μεταφορά του νοσοκού δικαίου στην Εθνική Νομοθεσία. Καταρχάς, καταφέραμε να ορίσουμε προτεραιότητες και να επικεντρωθούμε στις σημαντικότερες παραβιάσεις νοσιακού δικαίου. Έπειτα, Υπάρχουν κάποια ορόσημα πάνω στα οποία θα μπορέσουμε να ε, κάνουμε μια συγκριτική αξιολόγηση της εφαρμογής. Ε, υπάρχει διάλογος με τα κράτη-μέλη και επίσης προσπαθούμε να είμαστε σε άμεση επικοινωνία με τους ε, αρμόδιους φορείς και με τους πολίτες εν γέννη. Εκτιμούμε πολύ τις ε, προσπάθειες ε, του ελεκτικού συνεδρίου. Έχουμε σημειώσει όμως μεγάλη προσοχή τους τομείς όπου το ελεκτικό συνέδριο θεωρεί πως πρέπει να γίνουν περισσότερα. Ε, τον τρόπο καταρχάς με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι καταγγελίες των πολιτών. Ενώ είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι οι καταγγελίες είναι αναγκαίες έτσι ώστε να εντοπιστούν οι παραβιάσεις, από τις Βρυξέλλες είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουμε ε, την ε, ποιότητα αυτή των ε, καταγγελιών. Προσπαθούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε χρηστή διακυβέρνηση και να παρέχουμε καθοδήγηση και κατευθυντήριες γραμμές, να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες έτσι ώστε να κρίνουμε εάν χρειάζεται δράση. Επίσης προσπαθούμε να απαντούμε σε όλες τις καταγγελίες εντός 12 μηνών. Αντιμετωπίζουμε βέβαια πολλέ προκλήσει σχετικά με τη διαχείριση των καταγγελιών, διότι πολλέ φορέ οι καταγγελίε που φτάνουν στα χέρια μα ε, ε, λένε πράγματα ότι σα παρακαλώ αποζημιώστε με, σα παρακαλώ κάντε κάτι, διότι ε, έχουν παρεμβεί τα δικαιώματά μου. Το, τα, τα εθνικά δικαστήρια είναι αρμόδια για αυτό όμω. Οι πολίτε λοιπόν δεν έχουν αρκετή ενημέρωση έτσι ώστε να ξέρουν πού να απευθυνθούν. Έργο μας λοιπόν είναι να βοηθήσουμε τους πολίτε να βρουν τον κατάλληλο δίευλο επικοινωνία έτσι ώστε να, ε, να βρουν λύσει στα προβλήματά τους. Έπειτα, η διαφάνεια είναι ένα τομέα στον οποίο χρειάζεται βελτίωση. Έχουμε κάνει πάρα πολλά έτσι ώστε να βελτιώσουμε την διαφάνεια, όμως ε, πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα. Καταρχάς, οι πολίτες θέλουν να ξέρουν τι κάνουμε όταν ε, ασχολούμαστε με μία υπόθεση, όταν προσπαθούμε να επιβάλλουμε την νομοθεσία, πώς τη χειριζόμαστε. Αυτή την απέτηση προσπαθούμε να την ε, διαχειριστούμε δημοσιεύοντας εκθέσεις, ε, ανακοινώσεις για το ε, πώς αντιμετωπίζονται περιπτώσεις ε, παραβίασης του νοσιακού δικαίου. Επίσης, η δουλειά εδώ στην Επιτροπή σας είναι πάρα πολύ ε, χρήσιμη έτσι ώστε να γίνεται ο κατάλληλος έλεγχος και να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με, το, με τη δράση μας. Σε εθνικό επίπεδο, λοιπόν, προσπαθούμε και να συγκρίνουμε την εφαρμογή του νοσιακού δικαίου από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, έτσι ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πώς ακριβώ τα εθνικά του κοινοβούλια έχουν ε, μεταφέρει τις ε, οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εθνική νομοθεσία, αλλά και τι έχουν κάνει τα άλλα κράτη-μέλη. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Γι' αυτό και είναι απόλυτο αναγκαία συνεργασία με το Εθνικό Κοινοβούλιο, διότι εσεί είστε το πρώτο στάδιο Φυσικά πρέπει να η μεταφορά αυτή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας πρέπει να γίνεται ε, με τρόπο ομαλό, κατόπιν συζήτηση στα εθνικά κοινοβούλια, έτσι ώστε να τονιστεί η ευρωπαϊκή διάσταση της ε, πολιτικής που πρέπει να εφαρμοστεί. Θα ήθελα λοιπόν να ολοκληρώσω τονίζοντας ότι η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου είναι κοινό μας καθήκον και δεν είναι κάτι στατικό. Είναι κάτι που αλλάζει συνέχεια και προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε την ενωσιακή νομοθεσία. Ακριβώς διότι δεν πρέπει να είναι άκαμπτη. Πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια ανακοίνωση για την ενιαία αγορά, η οποία ανακοίνωση έγινε κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου, το οποίο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντοπίσει τους ε, τελευταίους φραγμούς για την ολοκλήρωση της ε, ενίας αγοράς. Εξετάσαμε τον ε, τομέα αυτό, βρήκαμε πως υπάρχει επίγουσα ανάγκη να τακτοποιηθούν νομικές εκκρεμότητες. Αυτό όμως που θεωρήσαμε πιο σημαντικό από όλα και θα το βρείτε με στην ανακοίνωση είναι ότι Εκεί που εντοπίστηκαν ελλείψεις ήταν στην ε, εφαρμογή σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω πως ε, μετά τη σημερινή έκρωση θα συνεισφέρουμε σημαντικά, ε, διότι χωρίς την ουσιαστική εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε. Προσβλέπω λοιπόν στην ανταλλαγή απόψεων και με χαρά μου θα ακούσω τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να δώσουμε το λόγο στην διαμεσολαβήτρια, την κυρία Μιλέη Ρέιλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι ανάμεσά σας για να συζητήσω ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να καταλάβουμε μερικές από τις δημοκρατικές προκλήσεις με τις οποίες βρισκόμαστε αντιμέτωποι. Η ικανότητα των ανθρώπων να καταλάβουν το πώς εφαρμόζονται οι νόμοι που επηρεάζουν την καθημερινή του ζωή είναι πεντουσία της δημοκρατίας. Είναι επίσης σημαντικό για μας, για την αυτονομία μας και για να μπορούμε να ελέγχουμε τον κόσμο. Να έχουμε δηλαδή την αίσθηση ότι μετράμε και ότι δεν καθορίζουν άλλοι το μέλλον μας σε μια διαρκώς παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και σε ένα κόσμο που οι νέες τεχνολογίες ασκούν ιδιαίτερα σημαντικό έλεγχο, δεν είναι εύκολο να, μπορεί, να πιστέψει κανείς, δεν είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς, ούτε εκείνοι ούτε τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να ελέγξουν τους νόμους που διέπουν τη ζωή μας. στο Brexit χρησιμοποιήθηκε το σύνθημα «Ξαναπάρτε πίσω τον έλεγχο» θεωρώντας ότι πραγματικά απευθύνεται σε μια βαθιά ψυχολογική ανάγκη πολλών ανθρώπων. Όταν οι άνθρωποι νιώθουν ότι έχουν χάσει τον έλεγχο, η αξιοπιστία και η νομιμότητα αρχίζουν να πάσχουν ακόμα και σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο. Το θέμα της απώλειας ελέγχου χρησιμοποιείται από τους ευρωσκεπτικιστές προκειμένου να πλήξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολλοί όμως Ευρωπαίοι πολιτικοί δημοσίως κατηγορούν τις Βρυξέλλες για νόμους ή πολιτικές εξελίξεις που γίνονται αντιληπτές με ανητικό τρόπο. Πολύ συχνά αυτό το κάνουν και όταν παίρνουν αποφάσεις για θέματα που μετά επικρίνουν ή δεν θέλουν να εφαρμόσουν. Αυτό είναι κάτι που προσπάθησα να αντιμετωπίσω μέσα από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πρόσφατα στην έρευνά μου για την λογοδοσία της διαδικασίας, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο, το δικαίωμα ενό Ευρωπαίου πολίτη να γνωρίζει τις απόψεις που υιοθετήθηκαν από την κυβέρνησή του δεν θα πρέπει να, να μειώνεται όταν η ίδια κυβέρνηση προτείνει εθνική νομοθεσία. Το, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διάφορους τρόπους για να ενημερώσει το κοινό σχετικά με το πώς αποφασίζονται οι νόμοι. Πέρσι ξεκίνησαν μια σειρά από διαδικασίες επί παραβάση. Αυτό βασιζόταν σε καταγγελίες από πολλούς αρμόδιους φορείς θα μπορούσαν να είναι και νομικές διαδικασίες. Για, ε, για να αναφέρουμε για παράδειγμα την οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία τους προκειμένου να επηρεάσουν την αλλαγή στους νόμους. Η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών είναι ένα άλλο σημαντικό εργαλείο το οποίο δεν έχει <clears throat> πλήρως εξελιχθεί. Το γραφείο μου και το γραφείο άλλων διαμεσολαβητών μπορούν να παίξουν ενεργό ρόλο. Είμαστε μια γέφυρα μεταξύ των πολιτών και της διοίκησης μέσω της συνεργασίας, μέσω του ε, ε, Ευρωπαϊκού Δίκτυου Διαμεσολαβητών. Προσπαθούμε να ρίξουμε μια γέφυρα με τους πολίτες ε, όταν τα προβλήματά τους έχουν μια ευρωπαϊκή διάσταση. Παράλληλα διεξάγουμε έρευνες στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει ένα θέμα εθνικής και ενωσιακής σημασίας. Όπως ξέρετε, η συνθήκη της Ρισαβόνας καθόρισε το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν έναν ε, συγκεκριμένο ρόλο να διαδραματίσουν, όπως για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των ε, της νομοθεσίας στο, ευρωπαϊκό, στο εθνικό δίκαιο. Ο διακοινοβουλευτικός διάλογος κατέστησε αυτό το ρόλο ακόμα πιο απτό και σήμερα ασχολούμεθα και με την εφαρμογή του νόμου, όχι μόνο με την νομοθεσία. Τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να μπορούν να ασκούν επιρροή και θα πρέπει να νιώθουν ότι μπορεί να διαδραματίσουν αυτό το ρόλο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Όταν οι πολίτες των Εθνικών Κοινοβουλίων προσπαθούν να επηρεάσουν τα πράγματα, οι προσπάθειές τους θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Τα κοινοβούλια θα πρέπει να ρίχνουν γέφυρες ανάμεσα στους πολίτες και θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως συγκεκριμένο παράδειγμα, θα ήθελα να πω ότι πέρα από τις αλλαγές που γίνονται στα πλαίσια της, ε, των μεταρρυθμίσεων, το πιο σημαντικό σημείο είναι το ε, κενό που υπάρχει ε, μεταξύ των προσδοκιών και των μέτρων που προτείνονται από την Επιτροπή. Αν κοιτάξουμε το θέμα, θέματα που αφορούν τα ύδατα, θα δούμε Πώς απήντησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εμπλεκόμενοι δυσαρεστήθηκαν ιδιαίτερα προκειμένου να έχουν κάποιο νόημα οι προσπάθειές τους. Εμείς θα πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις προσδοκίες των πολιτών ή των βουλευτών που θέλουν να καταβάλουν μια προσπάθεια να επηρεάσουν τα πράγματα. Θα πρέπει όμως να ξεκινήσουμε σε επίπεδο ευαισθητοποίησης. Θα πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν πώς μπορεί να ακουστεί η φωνή τους. Κοιτάζοντας προς τις ευρωπαϊκές εκλογές που πραγματικά θα αποτελέσει ένα σημείο αναφορά, συνειδητοποιούμε ότι αυτό είναι βασική προτεραιότητα. Θα πρέπει ο πολίτης να ξέρει ότι μπορεί να επηρεάσει τους νόμους όπου αποφασίζονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και πραγματικά περιμένω με ανυπομονησία να ενημερωθώ για το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης. Σας ευχαριστούμε. Μας ενέπνευσε ιδιαίτερος αυτή η εισαγωγή. Περνάμε στο πρώτο πάνελ τώρα της Δημόσιας Ακρόσης με θέμα τη μεταφορά, εφαρμογή και εκτέλεση του ενωσιακού δικαίου στα κράτη-μέλη. Και στο πρώτο τμήμα του πάνελ θα αναλύσουμε μερικές ε, ε, περιπτώσεις όπου μεταφορά και η εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών διατάξεων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των δύο επιτροπών ΠΕΤΗ και ΓΙΟΥΡΗ. Θα μιλήσουμε ε, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στα θέματα μεταφοράς στην τάξη και εφαρμογή. Και θα δούμε πώς μπορούμε να δυναμώσουμε τα εθνικά κοινοβούλια για να εξασφαλίσουν εμπρόθεσμη και σωστή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ε, ευρωπαϊκών ε, νομοθετικών διατάξεων. Και σίγουρα το, η πρώτη υπόθεση αφορά την οδηγία για τη διαμεσολάβηση που συνιστά ορόσημο γιατί πρόκειται για την πρώτη οδηγία που προβλέπει εναλλακτική επίλυση διαφορών σε θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου. Ε, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ευκολότερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη στα πλαίσια τη πολιτική μας να έχουμε έναν ευρωπαϊκό χώρο, ενιαίο χώρο δικαιοσύνη. και από αυτή την άποψη η οδηγία περί διαμεσολάβηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο που προωθεί μια κουλτούρα ε, όχι αντιδικίας ε, αλλά εναλλακτική επίλυση διαφορών, γιατί η διαμεσολάβηση διευρύνει την ε, πρόσβαση των πολιτών στα δικαστήρια, αποφεύγοντας χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες, ε, προωθώντας εναλλακτικού τρόπους επίλυση των διαφορών. Η διαμεσολάβηση έχει πολλά πλεονεκτήματα, χαμηλό κόστος, ε, σύντομο χρονικό διάστημα και εξυπηρετεί τις ανάγκες των ενδιαφερομένων. Και από την ε, έγκριση αυτής της οδηγίας, ε, η, οδηγία, η ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων έχει παρακολουθήσει τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, διοργανώνοντας σεμινάρια, ακροάσεις, συζητήσεις με πανεπιστημιακούς και μάλιστα πέρυσι υιοθετήσαμε και την έκθεση εφαρμογή για τις επιπτώσεις που έχει οδηγία περί διαμεσολάβησης στους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τη θέση ισχύ και η παρακολούθηση αυτού του θέματος ε, μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η οδηγία περί διαμεσολάβηση ήταν πολύ σημαντική γιατί αύξησε την επαγρύπνηση και την συνειδητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών για τα ωφέλη της διαμεσολάβησης. Αλλά η εφαρμογή της οδηγίας ε, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ως εκ τούτου έχουμε υποβάλει συστάσεις στα κράτη-μέλη προκειμένου να βαθμίσουν τις προσπάθειές τους, να εντείνουν την εφαρμογή τις οδηγίες αυτής ε, για τη διαμεσολάβηση στην, ε, στο εθνικό τους δίκαιο και θα ακούσουμε την παρουσίαση των επιμέρους υποθέσεων. Θα ήθελα να καλωσορίσω πρώτα την Μαρία Χωσέ Μαρτίνες ε, που είναι διευθύντρια σε θέματα νομικών υποθέσεων στη νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του νομικού συμβούλου του κυρίου Τρέξλερ, που βρίσκεται στο δικαστήριο, γι' αυτό κολλείεται σήμερα. Και λυπάται κυρίως ο νομικός σύμβουλος για την απουσία του, γιατί η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετείχε πολύ ενεργά σε αυτή την διοργάνωση και παρακολουθεί εκ του και σε αυτά τα θέματα. Σε μια κοινότητα δικαίου, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το θέμα της εφαρμογής του δικαίου βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Γιατί είναι η πεπτούσια του κράτους δικαίου. Και η ύπαρξη του δικαίου εξαρτάται από το σεβασμό των νομοθετικών διατάξεων και από την εφαρμογή του δικαίου. Και αν οι δημόσιε αρχέ δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα του νόμου, δεν υπάρχει κράτο δικαίου τελικά. Βέβαια, το ενωσιακό δίκαιο ε, είναι εκφύσεως ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του. Καταρχήν επειδή το ενωσιακό δίκαιο είναι ο καρπός ε, ενός διαλόγου μεταξύ 28, μεταξύ 28 διαφορετικών ε, ε, νομικών παραδόσεων και νομικής κουλτούρας και η διάρθρωσή του είναι αποκεντρωμένη. Δεν έχει, ουσιαστικό εκτελεστικό, δεν έχει ουσιαστική εκτελεστική εξουσία και χωρίς τα κράτη-μέλη την μέρημνα της εφαρμογής και της εξασφάλισης αποτελεσματικότητας του ενωσιακού δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι αφενός τα εθνικά κοινοβούλια εμπλέκονται στην μεταφορά του ενωσιακού δικαίου στην εσωτερική του ένωμη τάξη, όταν δεν έχουμε κανονισμούς που είναι αλλά οδηγίες, αλλά και οι διοικητικέ αρχές εμπλέκονται στη μεταφορά και στην εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Και μάλιστα σε ό,τι αφορά τη μεταφορά έχουμε κάποιες δυσκολίες. Καταρχήν ε, υπάρχει, υπάρχει διαφορά στη νομική κουλτούρα, στη νομική παράδοση. Αλλά υπάρχουν και διαφορετικές διαδικασίες ε, ε, εμπλοκής των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων και του βαθμού συμμετοχής των Εθνικών Κοινοβουλίων και των διοικητικών αρχών. Υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο που μας απασχόλησε πολύ τα τελευταία χρόνια. Το θέμα του κανονιστικού υπερθεματισμού, δηλαδή την προσθήκη ξένων στοιχείων εθνικών στο, στην ενωσιακή νομοθεσία στους κανόνες που είναι άμεσης εφαρμογής υπάρχει πιθανότητα διαφορετικών διοικητικών πρακτικών, διαφορετικής ε, νομικής ερμηνείας, οπότε το σύνολο του ενωσιακού δικαίου αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα ανομοιομορφίας. Δεν υπάρχει ομοιογένεια. Και η σημερινή ακρόαση θα μας επιτρέψει να εξετάσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, από τα παραδείγματα τέτοιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στην εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Τώρα, γιατί ε, θα πρέπει να ενδιαφέρεται ο νομοθέτης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει την εφαρμογή του δικαίου. Αλλά ασκείται κοινοβουλευτικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο έργο και τι δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των ενεργειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και για να βελτιωθεί η νομοθεσία, ο νομοθέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει ε, πώς διεκπεραιώνεται η όλη νομο... διαδικασία. Και η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτέλεσε το αντικείμενο της τελευταίας διοργανικής συμφωνίας για το ΕΦ νομοθετήν. Οπότε η και οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχονται να κριθούν για το αποτέλεσμα του νομοπαρασκευαστικού τους έργου. Οπότε είναι προφανές ότι και για το νομοθέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συνεργασία με τα υπόλοιπα κοινοβούλια, με τα εθνικά κοινοβούλια, είναι πολύ σημαντική. Λόγω του ρόλου που παίζουν τα εθνικά κοινοβούλια στη μεταφορά στην εθνική νομιτάξη, αλλά και λόγω του ε, εποπτικού τους ελέγχου στην εθνική εκτελεστική εξουσία. Αλλά σημαντικό ρόλο έχουν και οι εθνικοί διαμεσολαβητές, γιατί μπορούν να, να βρουν κάποια κοινά συμπτώματα σε ό,τι φορά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου κατά την εφαρμογή του στις εθνικές ένωμες τάξεις. Και θα ήθελα να προλάβω κάπως κάποια συμπεράσματα ή να προδικάσω κάποια συμπεράσματα της σημερινής ημέρας, γιατί νομίζω ότι το ζήτημα που θα πρέπει να μας προβληματίσει είναι κατά πόσο θα πρέπει να θεσμοθετήσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτή τη συνεργασία, τη διακοινοβουλευτική. Είτε μέσω συνεργασίας μεταξύ των διοικητικών δομών των εθνικών διαμεσολαβητικών φορέων, των εθνικών διαμεσολαβητών ή μέσω των διαφόρων πρωτοκόλλων που έχουν συμπεριληφθεί στη συνθήκη και προβλέπουν στο άρθρο 8 για παράδειγμα του πρώτου πρωτοκόλλου δυνατότητα δημιουργίας δομών μόνιμης κοινοβουλευτικής συνεργασίας. Έχουμε τέτοιο παράδειγμα με την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, με τα εξωτερικά θέματα ή με τη Europol. Οπότε υπάρχουν τέτοιε δομέ διοικητική συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Κοινοβούλων. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε κατά πόσο στο μέλλον θα πρέπει να θεσμοθετήσουμε και άλλα τέτοια επίπεδα συνεργασία. Σα ευχαριστώ, κυρία Ιγκλέσια, για τι προτάσει και τι συστάσει που θα μπορούσαν να μα καθοδηγήσουν οδηγήσουν καθ' τη διάρκεια της ημέρας. Περνάμε τώρα στη συζήτηση. Ε, μετά την ανάλυση της οδηγίας περί διαμεσολάβησης για εμπορικά και αστικά θέματα. Θα δώσω τώρα λόγο στον καθηγητή Τζουζέπε Ντεπάλο, που είναι καθηγητής ε, για το νόμο και την πράξη εναλλακτική επίλυση διαφορών στη νομική σχολή του Μίτσελ Χαμ Λάιν στο Σεντ Πολ των Ηνωμένων Πολιτειών. Για ένα τέταρτο. Έχει το λόγο. Tell Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως ε, βλέπετε, προτίμησα να πω κατευθείαν στο θέμα και να συνοψίσω ένα πολύ μεγάλο ενημερωτικό σημείο μας μέσα σε 15 λεπτά. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας ε, εξηγήσω γιατί κατά τη γνώμη μου η οδηγία δεν ε, έχει επιτύχει τους στόχους της είναι ε, βέβαια μια οδηγία ορόσημο, απέχει όμως πολύ από το να ε, γίνει αυτό το ορόσημο. Μάλιστα, σε ορισμένους κύκλους, η οδηγία του 2008 θεωρείται πως έχει προκαλέσει το εξής ε, περίεργο φαινόμενο. Καταρχάς, η διαμεσολάβηση είναι κάτι για το οποίο γίνεται λόγος και ακούγονται πολλά θετικά τα τελευταία 10 χρόνια, όμως μόνο το 1% όλων των ε, υποθέσεων ε, που καταλήγουν ε, σε, στα αστικά δικαστήρια ή εμπορικά δικαστήρια καταλήγουν σε διαμεσολάβηση. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει κάποια εγγύηση για μια εξισορροπημένη διαδικασία. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει ισορροπία ανάμεσα στην, ε, στις υποθέσεις που καταλήγουν στο δικαστήριο και σε αυτές που ε, περνάνε στα δύο διαμεσολάβησης. Το 2014 έγινε μία έρευνα που ποσοτικοποίησε ε, το κόστος της διαμεσολάβησης στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους ε, πολίτες. Η Επίτροπος Γιούροβα τότε, υπό την αιγύδα της Επιτρόπου Γιούροβα, το κόστος ανήλθε σε περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ ανά ε, έτος. Ανάμεσα σε 20 και 40, με συγχωρείτε. Το αστικό δικαστικό σύστημα δεν χρηματοδοτείται από τους ε, διαδίκους ε, και κατά μέσο όρο εκείνοι καταβάλουν μόνο το 25% του κόστους ο φορολογούμενος στην ουσία είναι εκείνος που ε, επιβαρύνεται με, το μεγαλύτερο κομμάτι του κόστους. Επίσης, ε, οι διάφορες διαφωνίες και συγκρούσεις είναι μια βιομηχανία που αναπτύσσεται συνεχόμενα. Σε έναν ολένα και πιο συνδεδεμένο κόσμο χρειάζεται οι επικοινωνίες να γίνουν πιο άμεσες έτσι ώστε να ε, συνδέουν τους ε, πολίτες σε όλον τον κόσμο. Αυτή η αμεσότητα όμως σημαίνει και περισσότερες διαφωνίες, οι καταλήγουν γρήγορα στο δικαστήριο ή στη βία. Πολλές φορές ε, δεν ε, γίνεται και απολύτως τίποτα. Η στη βια πολλε φορες αυτή το τιποτα η συγκρουση αντί να εισέλθουν ε, σε μία συζήτηση. Το περίεργο λοιπόν με την διαμεσολάβηση, αυτό το παράδοξο φαινόμενο έχει επιληθεί εν μέρη από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ περισσότερο από την Τουρκία. Η Ιταλία το 2015 είχε 15-20 φορές περισσότερες περιπτώσεις διαμεσολάβησης από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Και Φαίνεται ότι στις νέες υποθέσεις στις οποίες γίνεται διαμεσολάβηση ε, καταλήγουν σε επιτυχία. Ο αριθμός των υποθέσεων ε, μειώνεται κατά 30%. Ιδιαίτερα στον τομέα των ακινήτων, οι περιπτώσεις που καταλήγουν σε διαμεσολάβηση, σε διαμεσολάβηση στο 49%. Τώρα, περίπου το 85% των ε, υποθέσεων ε, δεν ε, καταλήγουν σε διαμεσολάβηση στην Ιταλία. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι Ιταλοί προτιμούν τη διαμεσολάβηση, αλλά ότι οι κανόνες εφαρμόστηκαν σωστά. Τώρα, στην Τουρκία, από, τα, από την αρχή του 2018 που υιοθετήθηκε το ιταλικό ε, μοντέλο έχουμε ένα ποσοστό επιτυχίας 67% των περιπτώσεων που κατέληξαν σε διαμεσολάβηση. Οι περιπτώσεις αυτές ε, είναι ε, από 13 έως 200.000 ανά έτος. Και έχουμε δει ότι υπάρχει μειωμένος αριθμός υποθέσεων που δεν καταλήγουν σε διαμεσολάβηση. Τι γίνεται λοιπόν, γιατί ε, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ο μηχανισμός διαμεσολάβησης χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου η ε, νομοθεσία ε, τον ευνοεί. Σε χώρες οι οποίες έχουν πολλές περιπτώσεις διαμεσολάβησης, γίνεται το αντίθετο. Υπάρχει ένας μηχανισμός opt-out. Ε, οι χώρε λοιπόν πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για να παροτρύνουν ε, τους ε, διαφωνούντες να καταλήξουν σε διαμεσολάβηση. Ο καλύτερος τρόπος ίσως να εξηγήσει κανείς ε, την ε, δύναμη ε, της διαμεσολάβησης και του μηχανισμού opt-out νομίζω πως φαίνεται από μία έρευνα του 2013 για τη διάσωση ανθρώπων και την περίπτωση δωρητών οργάνων. Η έρευνα αυτή κοίταξε τις περιπτώσεις συνένεσης των ε, δωρητών για να δοθούν ε, τα όργανα. Σε χώρες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό, η συνένεση ήταν ή ελάχιστη ή ε, η μέγιστη. Σε χώρες οι οποίες απαιτούν έγγραφη συνένεση, τα ποσοστά ήταν χαμηλά. Τι σημαίνει αυτό στη Γερμανία, α πούμε, πρέπει να υπογράψει ένα χαρτί που να λέει ρητά ότι ναι, συμφωνώ να ε, γίνω δωρητή οργάνων. Όταν ήρθε αυτή η ώρα όμω ελάχιστοι υπέγραψαν. Αυτές είναι οι χώρε αριστερά με το, την κίτρινη μπάρα. Στην γαλάζια μπάρα το κείμενο έλεγε ω εξή. Να υπογράψετε εάν δεν θέλετε να δωρηθούν τα όργανα σα σε άλλου. όσο λιγότεροι υπογράφουν, τόσο περισσότερα όργανα θα ε, διατεθούν σε άλλους ασθενείς. Η μέθοδος opt-out είναι πάρα πολύ σημαντική. Εάν αναλογιστεί κανείς πώς λαμβάνουν αποφάσεις ε, οι άνθρωποι. Το 2002 το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας δεν ε, απονεμήθηκε σε οικονομολόγο, αλλά σε ψυχολόγο, ο οποίος ε, διερεύνησε πώς ε, λειτουργεί ο ανθρώπινος νους ε, σε αβέβαιες συνθήκες. Προτιμήθηκε λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα, το, το κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Καλύτερα δηλαδή μια συμφωνία από πριν παρά να πάνε κάποιοι στο δικαστήριο με ένα βέβαιο αποτέλεσμα. Αυτό έχει να κάνει και με την έλλειψη ε, ελέγχου, αυτοελέγχου σε όλες τις επιτυχίες της ανθρώπινης ε, ζωής, ε, στην ε, σωστή διατροφή, στην διάσωση. Έχει αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι θα κάνουν το ασφαλέστερο. Όταν δηλαδή τους δίνει την δυνατότητα να, να κάνουν κάτι εθελοντικά ή να μην κάνουν κάτι εθελοντικά. Η λύση δεν θα πρέπει να είναι η παρότρινση, θα πρέπει να είναι η υποχρέωση να προβεί κάποιο η διαμεσολάβηση. Διαφορετικά δεν θα το κάνει. Και αυτή η έρευνα μας έδειξε και τις αδυναμίες της οδηγίας του 2008. Βλέπουμε στην οθόνη ότι υπάρχουν δύο άξονες. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι δεν παρέχεται μια δυνατότητα opt-out. μια, ε, υπάρχει μια δυνατότητα ενός ε, υποχρεωτικού μηχανισμού. Δεν ε, προβλέπονται βέβαια διάφορα στοιχεία, δεν αναγράφονται λεπτομέρειε. Δηλαδή, πόσο θα κρατήσει η διαμεσολάβηση, ποιο είναι υποχρεωμένο να πάει σε διαμεσολάβηση. Οι νομοθέτε πολλέ φορέ δεν ε, υπολόγισαν τις απρόβλεπτες ε, συνέπειες, την αιρεσιμότητα, την ε, προβλεψιμότητα, την κοινή λογική αρκετές φορές. Επίσης, υπήρχε εντύπωση ότι σε μια κουλτούρα διαμεσολάβησης, αυτή θα έχει και απήχηση στου πολίτε. Όμω αυτό ήταν λάθος σκέψη και λίγο πριν, μάλιστα, πολλά χρόνια πριν, ο, ο Βίδιος είχε πει ότι βλέπω το καλύτερο, αλλά ακολουθώ το χειρότερο. Οι άνθρωποι λοιπόν δεν πάνε αυθόρμητα στο σωστό. Και στη, γιατί αν το έκαναν αυτό, ούτε θα χρειαζόμασταν αστυνομία, ούτε φανάρια, ούτε νόμους, ούτε κανόνες ε, οδικής κυκλοφορίας. Τώρα, δύο χρόνια μετά την οδηγία, το δικαστήριο παρενέβη για να διορθώσει ορισμένα προβλήματα. Η περίπτωση Αλασίνη του 2010 ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πρώτον, αν θέλουμε το σύστημα να είναι αποτελεσματικό, δεν πρέπει να είναι opt-in, πρέπει να είναι opt-out. Αυτό ε, γράφει το δικαστήριο. Έπειτα, παρέχονται οι παράμετροι για να είναι επιτυχημένη μια διαμεσολάβηση, όμως ε, δεν είναι ε, υποχρεωτική, είναι προαιρετική. Και αυτό ήταν επίσης ένα πρόβλημα. Επίσης, η διαμεσολάβηση απεδείχθη αποτελεσματική σε ορισμένες περιπτώσεις Και το 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε τη δυνατότητα να αλλάξει το άρθρο 5.2 έτσι ώστε να συμπεριλάβει όλα τα θετικά στοιχεία. Δηλαδή ότι η διαμεσολάβηση πρέπει να γίνεται σε συνεργασία, ότι αν ε, η διαμεσολάβηση ξεκινήσει, τότε αναστέλλονται οι δικαστικές διαδικασίε. ότι η διαδικασία opt-out είναι εύκολη. Το 2017 το Κοινοβούλιο αποφάσισε να περιμένει και μάλιστα το 2016 είχε έρθει η ώρα για αναθεώρηση και αξιολόγηση τη οδηγία. Το 2017 όμως το Κοινοβούλιο αποφάσισε να μην αλλάξει ε, τίποτα στην οδηγία και να την αφήσει όπως ήταν. Με αυτή την απόφαση όμως οι εθνικοί νομοθέτες δεν γνώριζαν πώς ε, θα οριοθετήσουν μια επιτυχημένη διαμεσολάβηση και αντιμετώπισαν προβλήματα στο να θεσπίσουν νομοθεσία που θα είναι αποτελεσματική, με αποτελεσματικούς μηχανισμούς και στο ε, να θεσπίσουν μια νομοθεσία η οποία θα ανταπτύσσει αποκριθεί με επιτυχία στις ε, προκλήσεις και μάλιστα το ανώτατο δικαστήριο της Ρουμανίας έχει απορρίψει δύο φορές ε, υποθέσεις όπου ζητήθηκε να επιβληθεί υποχρεωτική διαμεσολάβηση. Πολλές φορές λοιπόν το δικαστήριο αποδυναμώνει μια ε, νομοθετική πρόταση και αυτό δεν είναι σίγουρα προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ε, αυτά προς το παρόν, η συνεισφορά των συνεργατών μου βρίσκεται στο τέλος της παρουσίασης. Κάποιοι από σας θα αναγνωρίσετε και το όνομά σας. Και θα ήθελα να πω στα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα προσπαθήσουν να επανεκλεγούν καλή τύχη και καλή τύχη σε εκείνους που θα ε, αποχωρήσουν. Ελπίζω την επόμενη φορά να ξαναβρεθούμε όχι για να συζητήσουμε τα προβλήματα της διαμεσολάβησης, αλλά για να γιορτάσουμε την επιτυχία της. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. για αυτά τα υποστηρικτικά λόγια που είπατε. Περνάμε τώρα στις ερωτήσεις από τους παριστάμενους. Όχι μόνο ερωτήσεις, δεχόμαστε σχόλια, παράθεση παραδειγμάτων, περιπτώσεων <clears throat> που πήγε καλά το θέμα της διαμεσολάβησης. I, I don't see, uh, comment. Η Μαρία τότε θα πάρει το λόγο. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Είπατε ότι ο νομοθέτης της Ένωσης δεν κατάφερε να δώσει ε, οδηγίες. Το θέμα όμως της διαμεσολάβησης ήταν ε, ιδιάζων. Όταν η Ένωση ξεκίνησε την όλη διαδικασία υιοθέτηση αυτής της οδηγίας, βεβαίως χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια. Ξεκίνησε η διαδικασία το 2000 με τη Λευκή Βίβλο λοιπά. Και νομίζω ότι τέθηκε σε εφαρμογή νομίζω το 2012. Τότε ολοκληρώθηκε η, περί... η περίοδος ε, μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Σε ορισμένες χώρες μέλη δεν υπήρχε η διαμεσολάβηση όταν υιοθετήθηκε η οδηγία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πήρε μια ομόφωνη απόφαση για αυτή την ομοθεσία γιατί υπήρχαν προβλήματα όπως το θέμα της επικουρικότητας γιατί η οδηγία περί διαμεσολάβησης βασίζεται στην εσωτερική αγορά, βασίστηκε από την αρχή και αυτό σημαίνει ότι εναρμονίζει κανείς πράγματα που δεν υπάρχουν. Μια ιδιαίτερα <clears throat> δύσκολη διαδικασία Ήθελα να κάνω αυτό το σχόλιο γιατί αυτό εξηγεί την έλλειψη ομοιογένειας καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ε, οδηγία η διαμεσολάβηση. Χρησιμοποίησα τη λέξη «απέτυχε» για να τραβήξω την προσοχή σας. Η διαδικασία ξεκίνησε το 1999 η πρόταση υποβλήθηκε το 2004, υιοθετήθηκε το 8. Είχα το προνόμιο να μιλήσω ενώπιόν σας το 2007, τη χρονιά πριν από την υιοθέτηση και επειδή ξεκίνησα τις διαμεσολαβήσεις, το 85 θεωρούσα ότι το ένα άρθρο δεν ήταν επαρκές. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα πήγαιναν καλά τα πράγματα. Ε, ε, πάρα πολλοί, ε, αναζητάνε ε, το καλύτερο, έτσι αντιμετώπιζαν τον νόμο περί διαμεσολάβησης. Όταν χρησιμοποίησα τον όρο απέτυχε, ήθελα να πω ότι στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ήταν ξεκάθαρο τι θα πήγαινε καλά και τι όχι. Στην Ιταλία υπήρχε νομοθεσία από το 93, στη Γαλλία το 94. Αυτό λοιπόν Λοιπόν που μπορούσε να δημιουργιαγήσει μια αγορά σε επίπεδο προσφοράς και ζήτησης ήταν γνωστό. Βεβαίως κανένας δεν είναι τέλειος συμπεριλαμβανομένου και αυτού του κοινοβουλίου. Αλλά από το 2008 μέχρι το 2018 το ε, <clears throat> κοινοβούλιο άρχισε το μελετάει το 11, μετά το 14, μετά το 16. Τότε κάνουμε τον απολογισμό μας αν ξεκινήσουμε από το Τάμπερε, ε, θα δούμε ότι είναι 19 χρόνια. Υπερβολικό θα έλεγα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είναι ο διακόπτης. Δεν είναι να αλλάξουμε τα μυαλά των ανθρώπων, είναι να κάνουμε τις σωστές νομοθετικές επιλογές. Η ομορφιά των νομοθετημάτων για τη διαμεσολάβηση είναι ότι προβλέπουν μία περίοδο δοκιμαστική. Δεν λένε ότι αυτό είναι οριστικό. Προβλέπεται περίοδος opt-in και opt-out. Σε ορισμένες ομοσπονδιακές χώρες, ε, η Αυστραλία για παράδειγμα, ε, υπάρχουν ε, ε περιοχές που έχουν ένα μοντέλο opt-in και άλλες που έχουν ε, το opt-out. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησα τον όρο «απέτυχε» παίρνω πίσω το 50% με έναν τρόπο διαμεσολάβησης. like, as, as you made an... Εξηγήσατε ε, αναφερόμενο στην ψυχολογία των πολιτών Μπορούμε να καταλάβουμε και την ψυχολογία των βουλευτών. Γιατί πήραν αυτή την απόφαση. Έχετε κάτι να πείτε. Νομίζω ναι. Ένας από τους συναδέλφους σας, όταν για πρώτη φορά μίλησε ενώπιον αυτού του ακροτηρίου πριν από πολλά χρόνια, αντί να χρησιμοποιήσω την έκφραση «απαιτούμενη», χρησιμοποίησα την έκφραση υποχρεωτική προσπάθεια. Ε, μου είπε λοιπόν αυτός ο βουλευτής, για μένα οτιδήποτε υποχρεωτικό είναι κακό. Πολλοί θεώρησαν ότι όρος υποχρεωτικό είναι κακό. Αν κοιτάξετε το άρθρο 2, φαίνεται ότι ενσταλάζει την ιδέα ότι ε, η απαιτούμενη διαμεσολάβηση είναι κακή. Ε, λέμε υπό τον όρο ότι δεν παραβιάζεται το δικαίωμα πρόσβαση σε προσφυγή στη δικαιοσύνη. Θεωρήθηκε δηλαδή η μεσολάβηση ένα ταμπού. Ένας συναδελφός μου από την ε, ε Ολλανδία αναφέρεται στην παρουσία φιλών, Μία φυλή υπέρ, μία φυλή κατά. Η πρόταση που είδατε στην ουσία θέτει σε εφαρμογή αυτά που λέμε. Είναι μια ε, μεσολάβη, διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο αυτών φυλών. Από την άλλη πλευρά αποδεικνύουμε ότι η, η μεσολάβηση σαν συστημα όπτιν δεν θα λειτουργήσει όπως δεν θα λειτουργήσει, δεν λειτουργήσε πουθενά. Αυτό δεν θα λειτουργήσει. Από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τους ανθρώπους. Ε, δεν κάνουμε αυτό, κάνουμε κάτι ενδιάμεσο. Προσπαθούμε να πείσουμε τους ανθρώπους να κάνουν μια προσπάθεια και ελέγχουμε μετά. Αυτό έχει ένα κόστος. Στο τέλος της χρονιάς πόσες περιπτώσεις έχουν ε, ρυθμιστεί, τι λένε οι άνθρωποι, τι λένε οι δικηγόροι. Οι δικηγόροι πολλές φορές ε, αντιτίθεται. Πολλές φορές ε, είχαμε απεργίες στην Αργεντινή, στην Ιταλία. Το νομικό επάγγελμα, ο νομικός κλάδος, τώρα είναι από τους πιο ένθερμους υποστηριχτές της ε, διαμεσολάβησης. Ο φόβος είναι ένα άλλο συνέστημα με το οποίο θα πρέπει να αναμετηθούμε, αλλά νομίζω ότι η προσοξεκτική εξήγηση το τι κάνουν οι άλλες χώρες ε, θα μας δώσει συγκεκριμένες ενδείξεις του τι μπορεί να εφαρμοστεί και τι όχι. Κουράγιο ε, λοιπόν και ενδεχομένως εξέταση και άλλων μοντέλων. Αυτός είναι ο δρόμος. Ε, δεν θα ήθελα να το μετατρέψουμε σε διάλογο με τον καθηγητή Ντεπάλο. Αλλά το θυμάμαι από το 2007 που είχαμε τις σχετικές συζητήσεις. Ε, εμένα δεν με σόκαρε ο όρος αποτυχία που χρησιμοποίησατε. Συμφωνώ μάλιστα με την ανάλυση σας. Γιατί γι' αυτό ακριβώς το λόγο στην οδηγία για τις ε, διαμεσολάβησεις έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς δεν εφαρμόζεται ε, σε όλα τα κράτη-μέλη με τον ίδιο τρόπο. Κάπως εφαρμόζεται, αλλά υπάρχουν τέτοιες διαφορές στην εφαρμογή, όπως είδαμε και από τις ε, διαφάνειές σας, καταδεικνύουν ακριβώς ότι δεν υπάρχει καμία ομοιομορφία. Υπάρχει παντελής ανομοιογένεια κατά την εφαρμογή αυτής της οδηγίας και δεν έχουμε καταφέρει να εναρμονίσουμε ή να εξασφαλίσουμε ίδιο επίπεδο εφαρμογή ή παρόμοιο επίπεδο εφαρμογή τη διαμεσολάβηση όλα τα κράτη-μέλη. Και αυτή είναι στην ουσία η κατάσταση. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ναι, ναι, συμφωνώ και μάλιστα θα έρθω σε αντίφαση με αυτά που είπα προηγουμένω. Γιατί ε, η Ιταλική νομοθεσία και η τουρκική νομοθεσία και η ελληνική νομοθεσία που τώρα βρίσκεται σε φάση αναστολής ε, ε, ακολουθεί το μοντέλο της οδηγίας. Αλλά δυστυχώς η οδηγία δίνει τόσο λίγες οδηγίες και είναι ασκεμένο το λογοπαίγνιο, είναι γιατί δίνει υπερβολική διακριτική ευχέρεια στους νομοθέτες. Μερικοί ήταν παράτολμοι, άλλοι άτολμοι. Δεν υπάρχουν όμως κοινά σημεία. Εμείς θέλαμε μια νομοθεσία που θα κατευθύνει καλύτερα τους νομοθέτες για το ποιο είναι σωστό να γίνει. Γι' αυτό μετά από 10 χρόνια εφαρμογή μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε αποτυχία. Βέβαια έχει αποδείξει κάποια αποτελεσματικότητα, αλλά χρειάστηκαν κάποια χρόνια. Ε, ο νόμος της τέλης του 2013 πέρασε μετά από μια διετία αμφισβήτησης ε, και συνταγματικής αμφισβήτησης. Τελικά βρέθηκε κάποια χρυσή τομή. Και αν ε, η διάταξη ήταν ε, με βάση την αρχική κατεύθυνση που σας έδωσα, δεν θα υπήρχε πρόβλημα ως προς τη συνταγματικότητα τουλάχιστον με βάση το δικαστήριο, γιατί θα είχε φανεί. Οπότε, αν η οδηγία έδινε περισσότερες οδηγίες, καθοδηγήσεις, θα είχε καλύτερο αντίκτυπο. Νομίζω ότι ως προς το συμπέρασμα συμφωνούμε. Μάλιστα. Αν δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο για σχόλια, πραγματικά θα με ενδιαφέρε η άποψη και των ε, συμμετεχόντων. Πώς βιώνουν τα κράτη-μέλη την ε, διαμεσολάβηση. Αλλά δεν βλέπω να θέλει κανείς το λόγο για να μας παραθέσει την εθνική του εμπειρία. Οπότε, μια και ολοκληρώσαμε το πρώτο πάρελ, θα πρότεινα μια σύντομη διακοπή πριν περάσουμε στο δεύτερο πάνελ που αφορά το περιβάλλον, τα δημόσια και, εθνικά, και ιδιωτικά σχέδια για το περιβάλλον και την εφαρμογή της οδηγίας του 2014. Ο κύριος ε, Πολσάκη έφυγε για να ψηφίσει σε μια άλλη επιτροπή, θα επιστρέψει σε ένα δεκάλεπτο και θα προεδρεύσει στο επόμενο πάνελ. Οπότε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. θα So, uh, Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε. Με ιδιαίτερη χαρά θα καλωσορίσω την κυρία Μάρτα Μπαγεστέρος. Ελπίζω να μην κατακρεώργησα το όνομά σας. Καλώς ήρθατε κυρία μου. Χαίρομαι που ήρθατε. Η κυρία Βαγεστέρος ε, είναι σύμβουλος ε, νομικών υποθέσεων και πολιτικής ε, και παροχή συμβουλών για τον νόμο και την πολιτική από το Law Policy Consulting στις Βρυξέλλες και ασχολείται με θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και ιδιωτικών και δημοσίων σχεδίων για το περιβάλλον. Αυτό θα είναι το θέμα του συγκεκριμένου πάνελ. Κύριε Βαγιστέρος, έχετε το λόγο. Δέκα λεπτά και λίγο παραπάνω δεν πειράζει. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να έρθω για να σας μιλήσω για την εφαρμογή της οδηγίας του 2014 για τη μελέτη αντικτύπου. Στόχος ε, της ε, ομιλία μου είναι να δώσω στο Κοινοβούλιο κάποια σημαντικά στοιχεία αυτής της οδηγίας του 2014 για την εκτεταμένη εκτίμηση αντικτύπου επιπτώσεων, στοιχεία που χρήζουν προσοχής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποια βασικά στοιχεία και στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Κυρίως γιατί η οδηγία παρόλο που τέθηκε σε ισχύ το 2014, θα πρέπει να μεταφερθεί από τα κράτη-μέλη στις εθνικές τους Ένωμες τάξεις το 2017. Ε, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τις νομοθετικές προτάσεις που τις έχουν κοινοποιήσει τα κράτη-μέλη και είναι σημαντικό και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου και της εφαρμογής ε, ε, και εκτέλεσης ε, του ενωσιακού δικαίου στα κράτη-μέλη θα πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεριμνήσει και να εξασφαλίσει την εφαρμογή, τη σωστή εφαρμογή στο εσωτερικό εθνικό δίκαιο των βασικών στοιχείων που θα σας παρουσιάσω σήμερα για την οδηγία αυτή. Επιπλέον, η οδηγία απαιτεί κάθε έξι χρόνια από το Μάιο του 2017 και μετά να υποβάλλονται εκθέσεις από τα κράτη-μέλη με την κοινοποίηση στοιχείων δεδομένων και πληροφοριών για το βαθμό εφαρμογής της οδηγίας. Δηλαδή τα κράτη-μέλη οφείλουν να συγκεντρώνουν πληροφορίες γιατί είναι υποχρεωμένα να παρέχουν ποσοτικά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πόσες μελέτες επιπτώσεων έχουν διενεργηθεί στα κράτη-μέλη, ε, να δώσουν πληροφορίες για το κόστος ε, της διεξαγωγής τέτοιων, τέτοιων εκτιμήσεων αντικτύπου και επίσης όλες αυτές οι εξολογήσεις αντικτύπου που έγιναν θα πρέπει να περιέχουν πληροφορίες που απαιτεί οδηγία για τέτοιου είδους εκτιμήσεις. Οπότε γι' αυτό το λόγο τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συγκεντρώνουν πληροφορίες συνεχώς. Δεν μπορούν να περιμένουν έξι χρόνια για να τις κοινοποιήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό λοιπόν και, το Εθνικό, και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φροντίσουν και να μεριμνήσουν στα κράτη-μέλη να αναπτύξουν τα απαραίτητα συστήματα για να μπορούν να συγκεντρώνουν τακτικά, σε αιτήσια βάση, σε τακτική βάση γενικώ, να συγκεντρώνουν τις πληροφορίες, ώστε να μπορούν σε αυτό το χρόνο και μέσα στην εξαιτία που απαιτεί η οδηγία να κοινοποιούν τα σχετικά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η οδηγία αυτή δεν είναι καινούρια. Ξεκίνησε το 1985 και πρωταρχικός της στόχος είναι η εξασφάλιση της συνεκτίμησης περιβαλλοντικών κριτηρίων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οπότε πριν δοθεί έγκριση για ένα δημόσιο ή ιδιωτικό σχέδιο για το περιβάλλον, θα πρέπει να γίνεται ανάλυση του αντικτύπου του σχεδίου αυτού για το περιβάλλον και θα πρέπει να γίνεται διεξοδική ανάλυση αυτών των επιπτώσεων. Αυτό το περιεχόμενο έχει οδηγία, δηλαδή πρωταρχικό τη στόχο είναι η περιβαλλοντική προστασία. Σημαίνει όμως και τη στιγμή που υιοθετήθηκε η οδηγία ο βασικός της στόχος ήταν να δηλώσει απερίφραστα ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν σημαίνει να διακοπούν όλα τα σχέδια τα αναπτυξιακά, αλλά θα πρέπει προηγουμένως να αναλυθούν οι επιπτώσεις αυτών των σχεδίων για το περιβάλλον. Προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια για μια βιώσιμη ανάπτυξη, για μια υφόρο ανάπτυξη. Η οδηγία έχει επικυρωποιηθεί πολλές φορές και η επικαιροποίηση αυτή έχει στόχο την προσαρμογή της οδηγίας στις τεχνολογικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, όταν υιοθετήθηκε η οδηγία για τη δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα ή όταν υιοθετήθηκε η Ιρλανδική συνθήκη για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του δημοσίου στη διαδικασία αυτή. Και κατά τα 25 χρόνια εφαρμογής της οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κάνει μια ανάλυση αυτής της εφαρμογής και να αναθεωρήσει την οδηγία. Γι' αυτό το 2012 πρότεινε μια νέα οδηγία που στόχο έχει την επίλυση κάποιων προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγηση της προηγούμενης οδηγίας. Δηλαδή, να μειωθεί η γραφειοκρατία, το διοικητικό άχθος ή να απλουστευτούν κάποιες διαδικασίες. Αυτά ήταν τα και οι αδυναμίες που βρέθηκαν στην αξιολόγηση ή ε, να ενισχυθούν οι στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που αποκτούν μεγαλύτερη σημασία τώρα δυνάμει των κλιματικών αλλαγών είναι της ανάγκης προστασίας της βιοπικιλότητας. Ποια είναι τώρα τα βασικά στοιχεία της οδηγίας που θα πρέπει να εξετάσουμε εν ώψη και της επόμενης κοινοβουλευτικής περίοδου. Καταρχήν θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η οδηγία αυτή είναι αρκετά διαδικαστική. Περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια. Τον έλεγχο, το screening, δηλαδή την διεξοδική εξέταση του σχεδίου, που είναι το αντικείμενο της ανάλυσης για την αξιολόγηση αντικτύπου, θα πρέπει να αποφασιστεί καταρχήν αν θα πρέπει ένα σχέδιο να υπαχθεί στη διαδικασία ε, μελέτης αντικτύπου. Και αυτό γίνεται με βάση αυτή τη διαδικασία του ελέγχου, του screening, ανάλογα με τη φύση, ε, την τοποθεσία ή τις διαστάσεις του σχεδίου. Αφού γίνει αυτή η πρώτη εξέταση και αποφασιστεί ένα σχέδιο να υπαχθεί στη διαδικασία αξιολόγησης επιπτώσεων, υπάρχει μια δεύτερη φάση όπου η αρμόδια αρχή αποφασίζει ποιο θα είναι το περιεχόμενο και το εύρος αυτής της μελέτης, της αξιολόγησης αντικτύπου. Και η τρίτη φάση είναι η υιοθέτηση της μελέτης περιβαλλοντικού αντικτύπου που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για το περιεχόμενο του σχεδίου, και το πώς επηρεάζει το περιβάλλον. Η οδηγία για πρώτη φορά ορίζει ποια είναι τα διάφορα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει η αξιολόγηση. Δηλαδή, τι πληροφορίες θα πρέπει να υποβάλει ο ανάδοχος του σχεδίου για να εξασφαλίσει τη σωστή διεξαγωγή της μελέτης αντικτύπου. Επίσης, τη διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί πέραν αυτών των τριών φάσεων που σας περιέγραψα. Για παράδειγμα, πώς γίνεται η προετοιμασία της αξιολόγησης αντικτύπου από τον ανάδοχο του σχεδίου με τις πληροφορίες που οφείλει να δώσει, τι διαβουλεύσεις θα πρέπει να γίνουν, τι εξέταση θα πρέπει να κάνει η αρμόδια αρχή και πώς θα εγκρίνει τα συμπεράσματα για την έκθεση αντικτύπου. Τι στοιχεία τώρα προτείνει η αναθεωρημένη οδηγία. Καταρχήν, ε, αναφέρει το εύρος των περιβαλλοντικών ε, παραγόντων που θα πρέπει να αναλυθούν. Αυτοί οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, αυτά τα περιβαλλοντικά στοιχεία που εξετάζονται, που είναι το αντικείμενο της αξιολόγησης, θα πρέπει να αναλυθούν ή να αξιολογηθούν με βάση το βασικό σενάριο. Και το βασικό αυτό σενάριο καθορίζεται και περιγράφεται καλύτερα στην αναθεωρημένη οδηγία, στη νέα οδηγία του 2014. Η οδηγία αυτή δίνει μια εικόνα του περιβάλλοντος, δηλαδή ποια είναι η παρούσα κατάσταση του περιβάλλοντος και ποιες είναι οι τάσεις για την περιβαλλοντική κατάσταση. Με βάση αυτό το στιγμιότυπο, αυτή την κατάσταση, γίνεται μια αξιολόγηση της διαδικασίας προκειμένου να αναβρεθεί κατά πόσο οι επιπτώσει για το περιβάλλον θα είναι περιβαλλοντικοί παράγοντε θα αναλυθούν, για παράδειγμα, ή όχι. Ποιοι ε, περιβαλλοντικοί παραγοντε θα αναλυθούν. Για παράδειγμα, κατάσταση του ύδατο, ε, του εδάφους, ε, του αέρα. Αυτό περιλαμβανόταν και στην προηγούμενη οδηγία. Αλλά η νέα οδηγία, η αναθεωρημένη οδηγία, προσθέτει και την ανάγκη εξέτασης των επιπτώσεων και στις κλιματικές αλλαγές. Και στο παράρτημα 4 της οδηγίας αναφέρεται ότι αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορά το μετριασμό των κλιματικών αλλαγών, δηλαδή τις ε, εκπομπές αερίων στην ατμόσφαιρα, αλλά και τους παράγοντες προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές. Αυτά είναι τα νέα στοιχεία που προσθέτει η αναθεωρημένη οδηγία. Επίσης, η οδηγία τονίζει την ανάγκη εξέτασης ε, των επιπτώσεων του σχεδίου από τη σκοπιά της βιοπικιλότητας. Και η βιοπικιλότητα ορίζεται ως ε, τα ενδιατήματα και ε, τα είδη που τη χάνουν προστασίες δυνάμει της οδηγίας για τη φύση. Natura 2000. Και επίσης άλλος στόχος της οδηγίας είναι να εξασφαλίσει μία συνέπεια και μία συνοχή με τα άλλα νομοθετήματα της, οδη... της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, οδηγίες προστασίας της φύσης επίσης απαιτούν κατάλληλη αξιολόγηση αντικτύπου των σχεδίων που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στη βιοπικιλότητα ενδιατημάτων και ειδών χλωρίδας και πανίδας. Και είναι δύσκολο για έναν ανάδοχο σχεδίου να έχει την υποχρέωση να εκπονήσει μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου και μελέτη αντικτύπου ε, από τη σκοπιά των οδηγιών για την προστασία της φύσης. Οπότε η νέα οδηγία προσπαθεί να καταστήσει πιο αποτελεσματική τη διαδικασία και να απαιτεί μόνο μία ενιαία διαδικασία μελέτης για τον αντίκτυπο του σχεδίου στη βιοπικιλότητα. Η οδηγία για την μελέτη αντικτύπου, περιβαλλοντικού αντικτύπου είναι ευρύτερη από την οδηγία αντικτύπου για τη φύση και εξετάζει τις επιπτώσεις του σχεδίου για τη βιοπικιλότητα όχι μόνο σε οικοσυστήματα και διαιτήματα που τη χάνουν προστασίες με βάση το Natura 2000, έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογή η μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου, αλλά το βασικό της στοιχείο είναι να εξασφαλίσει ότι χάρη σε αυτή τη συντονισμένη διαδικασία που προβλέπει μία και μόνο εκτίμηση, να έχουμε μια τέτοια βελτιωμένη έκθεση αντικτύπου, μια βελτιωμένη μελέτη αντικτύπου. Αυτός είναι ο στόχος της οδηγίας. Και από αυτή την άποψη η ανάλυση του βασικού σεναρίου είναι παρόμοια και καθορίζεται διεξοδικά σε κάποια καθοδηγητικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμπερίληψη της βιοπικιλότητας στην οδηγία για τη μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Και πρόσφατη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκπονήσει και κάποιες κατευθυντήρες γραμμές για την οδηγία του 2014 για την μελέτη αντικτύπου για το περιβάλλον. Εκεί προτείνονται διάφορες μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό του βασικού σεναρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλο στοιχείο που απαιτεί οδηγία είναι στην αξιολόγηση επιπτώσεων να συμπεριληφθούν και τα σορευτικά αποτελέσματα που θα έχει το σχέδιο στο περιβάλλον. Σορευτικές επιπτώσεις. Στις προηγούμενες εκδοχές της οδηγίας, ένα από τα βασικά προβλήματα που εντοπίστηκαν ήταν ότι πολλά σχέδια είχαν ε, κατατεμαχιστεί σε μικρότερα για να αποφύγουν την υποχρέωση ε, διεξαγωγής μελέτης επιπτώσεων. Όταν έχουμε πιο μικρή εμβέλεια σχέδια, παρακάμπτεται η υποχρέωση εκπόνησης ε, αξιολόγηση αντικτύπου. Και αυτό το πρόβλημα ήταν το δικείμενο πολλών αναφορών και πολλών καταγγελιών και και μάλιστα ε, οδήγησε στην παραγωγή αρκετής νομολογίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γιατί το δικαστήριο επέμεινε στο γεγονός ότι έπρεπε να γίνει ανάλυση όλων των ε, σχεδίων ε, που εκπονώνταν σε μια περιοχή και που θα είχαν σορευτικές επιπτώσεις στην περιοχή αυτή και μιλούσε όχι μόνο για τα τρέχοντα σχέδια αλλά και για τα μελλοντικά σχέδια. Είχαμε πρόσφατη απόφαση στην Ιταλία όπου το δικαστήριο επέμεινε ότι η υποχρέωση δεν αφορά μόνο τα υπάρχοντα σχέδια αλλά και τα μελλοντικά ως προς τις επιπτώσεις που θα έχουν σε συγκεκριμένη περιοχή. Οπότε η τελευταία εκδοχή της οδηγίας τονίζει την ανάγκη ανάλυσης των σωρευτικών επιπτώσεων όλων των σχεδίων, των συναφών σχεδίων σε μια περιοχή. Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να εξεταστεί στο μέλλον είναι το γεγονός ότι η οδηγία απαιτεί περιγραφή και όλων των λογικών εναλλακτικών λύσεων που έχουν εκτιμηθεί. Όχι μόνο των εναλλακτικών λύσεων, αλλά και των λόγων για, το, για τους οποίους επιλέγει η συγκεκριμένη λύση και επίσης ε, ζητά και μια συγκριτική ανάλυση των επιπτώσεων των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων στο περιβάλλον. Ένα πρόβλημα άλλο που εντοπίστηκε επ' ευκαιρία της αναθεώρησης οδηγίας είναι ότι η απόφαση των αρμοδίων αρχών να εγκρίνει να απορρίψει ε, ένα σχέδιο στην απόφαση αυτή να υπάρχει περιγραφή των μέτρων που θα έπρεπε ε, να εφαρμόσει ο ανάδοχος του σχεδίου, ώστε να αποτρέψει, να προλάβει, να μειώσει ή να αντισταθμίσει τα αποτελέσματα στο περιβάλλον, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Υπήρχε απόφαση και κάποια προφανή μέτρα, αλλά δεν ακολουθούσε ένας μηχανισμός ελεγκτικός για να εξακριβωθεί κατά πόσο ο ανάδοχος όντως είχε ε, εφαρμόσει αυτά τα μέτρα που πρότεινε η αρμόδια αρχή στην απόφασή της. Με την οδηγία προβλέπεται πια υποχρέωση να, προσδιοριστούν τα μέτρα παρακολούθησης και άρα και ένας μηχανισμός παρακολούθησης που θα έπρεπε να θεσπίζεται στην ίδια την απόφαση, να αναφέρονται οι παράμετροι ε, για τον έλεγχο του σχεδίου και η διάρκεια των ελεγκτικών μέτρων. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της οδηγίας. Και μάλιστα έτσι εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της οδηγίας για την αξιολόγηση του αντικτύπου. Ένα άλλο στοιχείο επίση πολύ σημαντικό της οδηγίας για τη μελέτη αντικτύπου και της διαδικασία είναι η δημόσια συμμετοχή, η συμμετοχή του δημοσίου. Η οδηγία ενισχύει την ανάγκη της συμμετοχής του δημοσίου και μιλά για την αποτελεσματική συμμετοχή του δημοσίου. Πριν τη χορήγηση της έγκρισης του σχεδίου, η οδηγία απαιτεί να ενημερώνεται το κοινό και μάλιστα η οδηγία αναφέρεται σε όλες τις πληροφορίες που θα πρέπει να κοινοποιούνται ώστε να γνωρίζει το κοινό και να έχει την ευκαιρία να ε, αντιδράσει το σχέδιο ή να εκφράσει τις ανησυχίες του για το σχέδιο. Και επίσης απαιτεί πληροφορίες αυτές να παρατίθενται ηλεκτρονικά, είτε δηλαδή στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής, που είναι αρμόδια με τη λήψη της απόφασης. Εξασφαλίζεται λοιπόν η δημόσια συμμετοχή. Επίσης, η οδηγία απαιτεί μετά τη λήψη της απόφασης να δημοσιεύονται οι πληροφορίες. Δηλαδή, οι πληροφορίες η απόφαση θα πρέπει να δημοσιοποιείται. Και επίσης, να αναφέρονται και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια της διαβούλευσης και πόσο ελήφθησαν υπόψη ανησυχίες του κοινού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ήδη είχε ζητήσει να δίνονται αυτές οι πληροφορίες. Μόνο όμως μετά από αίτημα των πολιτών ή του, των ενδιαφερομένων. Ενώ η οδηγία είναι ακόμη πιο φιλόδοξη και απαιτεί οι πληροφορίες αυτές να παρέχονται αυτόματα δημόσια, χωρίς να χρειάζεται συγκεκριμένο αίτημα για την παροχή τους. Τώρα, τι γίνεται σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή, τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Το Μάιο του 2017 τα κράτη-μέλη πρέπει να ε, μεταφέρουν ε, στην νομοθεσία τους την οδηγία, εγκρίνοντας τις οικίες νομοθετικές διατάξεις. Από πληροφορίες που έχουμε γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία σε επιπαρεβάση για εκπρόθεσμη μεταφορά και εκπρόθεσμη κοινοποίηση της εθνικής νομοθεσίας που μεταφέρει ε, την ε, σχετική οδηγία ε, και ασκήθηκαν τέτοιε διαδικασίε επί σε 21 χώρε. Κατά 21, 21 χώρε σε σχέση με τι 28 Επίσης, με βάση τη Συνδική για τη Λειτουργία για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ε, δίνεται δυνατότητα στο δικαστήριο να επιδικάσει πρόστιμα για εκπρόθεσμη μεταφορά χωρίς προηγούμενη άλλη ε, έκδοση απόφασης. Βέβαια τα κράτη-μέλη ήδη κοινοποιούν τις, τα νομοθετικά τους μέτρα και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το κατά πόσο η οδηγία έχει μεταφερθεί σωστά στα εθνικά δίκαια. Και αυτή η εξέταση γίνεται εν μέρει και από τη δική μου εταιρεία. Η οδηγία για την αξιολόγηση αντικτύπου παρόλο που τέθηκε σε ισχύ το 2014, στην ουσία θα έχει αντίκτυπο, δηλαδή θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2017, γιατί τότε θα ενσωματωθεί στα εθνικά δίκαια. Και γνωρίζουμε από πληροφορίες που έχουμε λάβει τι νομοθετικά μέτρα θα υιοθετήσουν τα κράτη-μέλη για να μεταφέρουν την οδηγία. Χώρες όπως η Ιρλανδία έχουν παρουσιάσει πολύ καλές πρακτικές. Εκεί ήδη έχουμε κάποια στοιχεία για το τι μορφή θα έχουν τα σχετικά νομοσχέδια. Γιατί ε, έγιναν δημόσιες διαβουλεύσεις ε, και δόθηκαν πληροφορίες. Και στη Γαλλία το Συμβούλιο Επικράτης είπε ότι ήδη παρουσιάστηκαν κάποιες παραβιάσεις της οδηγίας ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υποχρέωση παροχής πληροφοριών ή την ε, αποφυγή σύγκρουσης αρμοδιοτήτων ε, ή συμφερόντων μεταξύ των ε, αρμόδιων αρχών που λαμβάνουν την απόφαση για την έγκριση ενός σχεδίου. Ε, πολλές φορές συμπίπτουν με τους αναδόχους των σχεδίων. Ήδη λοιπόν έχουν εντοπιστεί κάποια προβλήματα αντίστοιχα με αυτά των προηγούμενων οδηγιών. που προσπαθεί να λύσει η νέα οδηγία. Είναι σημαντικό λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια να μεριμνήσουν ώστε όλα αυτά τα στοιχεία της νέας αναθεωρημένης οδηγίας ε, να ληφθούν υπόψη κατά τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τώρα. Η οδηγία ε, ήταν το δικείμενο αριθμών καταγγελιών και ε, αιτιάσεων. 12% των διαδικασιών επί παραβάση αφορούσαν την οδηγία για τη μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Το 2017, το 2016 μάλλον, είχαμε 70 αναφορές από τις 314 γενικώ αναφορές που αφορούσαν τη συγκεκριμένη οδηγία. Οπότε είναι αρκετά τα υψηλά τα Το 2016, συγγνώμη, 70 από τις 348 νέες ε, καταγγελίες αφορούσαν ε, το περιβαλλοντικό δίκαιο και τη νέα οδηγία. Οπότε θα πρέπει να συμπληρωθούν οι κατευθυντήρε γραμμές, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εφαρμοστεί η νέα οδηγία. Βρισκόμαστε σε πολύ πρώιμη φάση ακόμη. Γνωρίζουμε όμως ότι κάποια στοιχεία της οδηγίας ίσως δημιουργήσουν προβλήματα στο μέλλον. Για παράδειγμα, η έννοια της βαρύτητας, της σημαντικότητας, συγκνήφικας. τι σημαίνει ότι ένα σχέδιο θα έχει σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον, γιατί η οδηγία δεν προσδιορίζει αυτή την έννοια της βαρύτητας, το πόσο σημαντικό θα είναι το σχέδιο. Η, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει κάποιες κατευθυντήρες γραμμές στα κράτη-μέλη για το τι σημαίνει βαρύτητα, με βάση το βασικό σενάριο και τι σημαίνει ως προς τη μεθοδολογία να εκτιμηθεί κατά πόσο ένα σχέδιο θα έχει σημαντικό αντίκτυπο. Και γι' αυτό προτείνεται να προσδιοριστεί μια μεθοδολογία. Για παράδειγμα υπάρχει ένα σχέδιο, το σχέδιο Imperia, που προτείνει μια μεθοδολογία παρόμοια με το εργαλείο RV, με βάση το Excel και δίνει ένα εργαλείο για να αξιολογείται η βαρύτητα ενός σχεδίου και να γίνεται μια σύγκριση των εναλλακτικών λύσεων για το σχέδιο αυτό, προκειμένου να γίνει δυνατή μια σωστή ανάλυση, μια άρτη ανάλυση και αξιολόγηση του αντικτύπου. Κάποια συμπεράσματα τώρα. Θα θέλαμε να παρατηρήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια να εξασφαλίσουν ε, κατάλληλο έλεγχο της εφαρμογής της οδηγίας υπό το πρίσμα όλων αυτών των στοιχείων που σας ανέφερα και να εξασφαλίσουν σωστή μεταφορά και εφαρμογή όλων αυτών των στοιχείων της νέας οδηγίας. Αυτά και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω στις απορίες σας. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και επαγγελματική ανάλυση που κάνατε, διότι πράγματι εντοπίστηκαν κάποια σοβαρά προβλήματα και αυτή είναι μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις χώρες αυτές. Υπάρχουν 21 κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν διαδικασίες σε παραβάση. Αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ε, κρατών μελών και νομίζω πως είναι καλό να σταλεί ένα μήνυμα. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε και για τις συστάσεις που κάνατε. Τώρα κυρίες και κύριοι θα ανοίξει η συζήτηση, αν έχετε σχόλια, ερωτήσεις για τους ε, προσκεκλημένους ε, μας, την προσκεκλημένη μας, έχει έρθει η ώρα να τις κάνετε. Έχω όμως ε, ενημερωθεί ότι ο David Law, πρώην μέλος της Επιτροπής Αναφορών, έχει έρθει και έχει ζητήσει το λόγο. Και ο κύριος Λαπτή, την Επιτροπή ανάπτυξη, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ξέρω πως ε, δεν έχουν δικαίωμα τα μη μέλη να συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις. Ευχαριστώ όμως πάρα πολύ. Πράγματι πρέπει να δούμε πως είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι είναι ανάγκη να θεωρηθεί η οδηγία και αυτό συνέβη ακριβώς διότι οι αναφορές που ε, έστειλαν οι πολίτες πολλών χωρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαν ε, να κάνουν φυσικά με αυτήν την αναθεώρηση της οδηγίας. Αυτό που μόλις ακούσαμε, την παρουσίαση δηλαδή της ε, κυρίας Μπαλεστέρας, αφορά πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Στην Επιτροπή Αναφορών προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει των πολιτών και μάλιστα ένα μέλος της Επιτροπής Αναφορών, ο κύριος Χουντής, ήταν εισηγητή της έκθεσης, η οποία τόνιζε ακριβώς αυτά τα κενά που υπήρχαν ανάμεσα στην προηγούμενη και, σε, στην επόμενη οδηγία και αυτές τις ε, αλλαγέ. Χρειάζεται λοιπόν να ενισχυθούν τα δικαιώματα των πολιτών και νομίζω πως ε, δεν είναι τυχαίο ότι η συγκεκριμένη οδηγία επιλέχθηκε. Διότι νομίζω πως ε, με αυτήν την οδηγία φαίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η φωνή των ε, πολιτών και σε αυτή την περίπτωση συνεργάστηκε πολύ καλά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να εγκριθεί αυτή η αναθεώρηση. Ωστόσο, όπως είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια, εκκρεμούν ακόμα διάφορα προβλήματα. Και αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι χρειάζεται τόσο πολύ καιρό έτσι ώστε να εγκριθεί η αναθεώρηση της οδηγίας, η οποία έγινε πριν από δύο χρόνια. Και πως οι περιπτώσεις ε, διαδικασίες παραβάσεις νομίζω φανερώνουν ακριβώς αυτό. Υπάρχει λοιπόν ένας δισταγμός ε, στα κράτη-μέλη για να αναλάβουν δράση και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την οδηγία προς όφελος όχι μόνο των πολιτών και των ε, τοπικών κοινοτήτων που τις αφορά ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος ορισμένων έργων υποδομής, ε, αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένα παραδείγματα. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα έργο το οποίο συζητάει η Επιτροπή Αναφορών πάρα πολλά χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε πως ε, πρόκειται για ξεκάθαρη περίπτωση παραβίασης ε, της οδηγίας για τα ενδιαιτήματα. Ακόμα λοιπόν προσπαθούν οι αρχές να αντιμετωπίσουν αυτές τις ε, κατάφορες παραβιάσεις της ε, νοσιακής ε, νομοθεσίας. Και νομίζω λοιπόν πως αυτό είναι μία απόδειξη του τι συμβαίνει και θα βοηθούσε πολύ εάν φτάνουν συχνά τέτοιες περιπτώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι χρειάζεται να συνεργαστούμε με την Κομισιόν και με τα κρατημέλη για να επιληθούν αυτά τα σοβαρά προβλήματα. Πολύ συχνά εμφανίζονται καταγγελίες όταν πρόκειται για τεράστια έργα υποδομών ε, και υπάρχουν πολλά συμφέροντα πίσω από αυτά τα έργα, κατασκευαστικές εταιρείες, διάφοροι φορείς ε, κτλ. Υπάρχουν λοιπόν ε, πολλά συμφέροντα, πολλά κονδύλια και αυτό έχει εμποδίσει, αποθαρρύνει τους πολίτες να οργανωθούν και να αντιδράσουν. Πολλές φορές μάλιστα ε, τους έχει αποθαρρύνει αρκετά επιθετικά. Είναι λοιπόν σημαντικό τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση για να προστατεύσουν τους Ευρωπαίους πολίτες και το περιβάλλον. Για παράδειγμα, ε, σε ό,τι αφορά τους στόχους για την βιοπικιλότητα, για την ε, οδηγία, για τα πουλιά και τα ενδιατήματά τους, Όμως για να συμβεί αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι πιο μαχητική. και να φέρει τα κράτη-μέλη που παραβιάζουν το, το ενωσιακό δίκαιο ενώπιον του δικαστηρίου, γιατί πρέπει να λογοδοτήσουν. Σίγουρα υπάρχουν πολλές ευθύνες στην ίδια την Κομισιόν και στους αρμόδιους επιτρόπους για την αποτελεσματική ε, εφαρμογή τη νομοθεσία. Όμω η καλύτερη λύση είναι η συνεργασία. Συνεργασία με τα κράτη-μέλη, με τα κοινοβούλια των κρατών μελών, έτσι ώστε να ε, διασφαλιστεί ότι όταν ε, γίνονται τόσε προσπάθειε και από του πολίτε και από το κοινοβούλιο για να αναθεωρηθεί η νομοθεσία, αυτό πρέπει να εφαρμόζεται αποτελεσματικά επιτόπου. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στον επόμενο ε, ομιλητή. Κάποιος, ε, κάποια ερώτηση, σχόλιο, παρακαλώ εσείς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω μία ερώτηση προς ε, την προσκεκλημένη σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων και πώς αυτό αντιμετωπίζεται στην οδηγία συμφωνώ και με την παρουσίαση και με τον ε, κύριο Λό, ο οποίος ε, είπε ότι οι περισσότερες καταγγελίες ε, αφορούν ακριβώς αυτήν την οδηγία. Και νομίζω πως αυτή η οδηγία είναι εξαιρετικά σημαντική, ακριβώς γιατί επιτρέπει στους πολίτες να καταφύγουν σε ένδυκα μέσα χρησιμοποιώντας μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ προβλήματα τα οποία διαφορετικά θα ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Για παράδειγμα, η χορήγηση ε, αδειών για διάφορα έργα. Ιδιαίτερα για τα πολύ μεγάλα έργα όπου δημιουργούνται διάφορα ζητήματα και μεγάλη ανησυχία στους πολίτες. Και η οδηγία αυτή είναι ο μόνος ε, σύνδεσμος των πολιτών και η μόνη δυνατότητα να βρουν κάποια βοήθεια, κάποια συνδρομή εκτός εθνικού επίπεδου. Γι' αυτό λοιπόν ε, περνάω σύντομα στην ερώτησή μου. Πολύ συχνά βλέπουμε ότι οι εκτιμήσεις περιβαλλοντικού αντικτύπου πολύ συχνά οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων κατά την ε, κατάρτιση της ίδιας της ε, μελέτης αυτής. Δηλαδή, αυτό που υποτίθεται πως είναι μία αξιολόγηση αμερόληπτη και επαγγελματική η οποία εξετάζει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο ενός ε, πολύ μεγάλου έργου πολύ συχνά καταλήγει να δικαιολογεί και να επιχειρηματολογεί υπέρ της ε, δημιουργίας και της κατασκευής αυτού του έργου. Πολύ συχνά λοιπόν βλέπουμε ότι αυτές οι εκτιμήσεις περιβαλλοντικού αντικτύπου ε, λένε ότι το καλύτερο μπορεί να συμβεί στο περιβάλλον είναι να ε, χτιστεί αυτό το τεράστιο έργο μέσα σε ένα δάσος παρθένο. Και φυσικά, αν ψάξει κανείς λίγο πιο μέσα, θα δει ότι αυτές οι εκτιμήσεις περιβαλλοντικού αντικτύπου έχουν χρηματοδοτηθεί από μεγάλους ομίλους κατασκευαστικούς. Γι' αυτό λοιπόν η ερώτησή μου προς την Επιτροπή έχει ω εξή. Τι γίνεται με τη σύγκρουση συμφερόντων, υπάρχει κάτι τέτοιο στην οδηγία, διότι αυτό ακριβώ το στοιχείο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στην εφαρμογή μια ε, οδηγίας ε, και ιδιαίτερα στην περίπτωση του περιβάλλοντος αυτό μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο η τελευταία παρέμβαση ήταν από τον κύριο Μποζούρτη από τη Μάλτα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει κάποια άλλη παρατήρηση, κάποια άλλη ερώτηση που θα θέλετε να θέσετε, παρακαλώ. Θα ήθελα να πάρω το λόγο κάνοντας μία ερώτηση. με μέλος του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση στην εισηγήτρια ως προς τον ορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο ολοκληρωμένη αξιολόγηση ενός προγράμματος τι σημαίνει μία μακρόπνοη εξέταση των εξελίξεων σε μια περιοχή. Γιατί πάρα πολύ συχνά προκύπτει μια σύγκρουση όταν διαχωρίζεται η γενική αξιολόγηση από μια αξιολόγηση που επικεντρώνεται στο περιβάλλον. Όταν έχουμε να κάνουμε με ένα νέο έργο. Η δεύτερη ερώτηση. Με τι τρόπο η οδηγία εμπλέκει διάφορα, συμπεριλαμβάνει διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, τοπικής, εθνικής, περιφερειακής, εθνικής, σε ό,τι αφορά τι διαδικασίε ελέγχου και παρακολούθησης του ίδιου του έργου, αλλά και της μελλοντικής διαχείρισης του ελέγχου σε επίπεδο διαχείρισης του ίδιου του έργου. Ευχαριστώ. κυρία Μανουέλα Ρωσίνη από την Ιταλία. Επόμενη παρατήρηση. Ερώτηση. Αν δεν κάνω λάθος, δεν θέλετε να κάνετε άλλες ερωτήσεις, παρακαλώ. Παρακαλώ, να δώσουμε το λόγο στην ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την πρώτη ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Υπάρχει ένα νέο άρθρο στην οδηγία, το 9α, το οποίο προβλέπει ότι σε φυσιολογικές περιπτώσεις υπάρχει υποχρέωση που προκύπτει από την οδηγία ο ανάδοχος του σχεδίου να δώσει πληροφορίες και αξιολόγηση. Μετά τις πληροφορίες αυτές τις συγκεντρώνουν οι αρμόδιες αρχές, τις αναλύουν, αναλύονται οι πληροφορίες δηλαδή, αναλύονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβουλεύσεων και λαμβάνουν αποφάσεις. Όταν ο ανάδοχος είναι ο ίδιος με την αρμόδια αρχή, προκύπτει ένα πρόβλημα και αυτό είναι κάτι που έχει οδηγήσει σε πολλές καταγγελίες. Αυτό που λέει αυτό το άρθρο είναι εκεί που η ανάδοχος αρχή ε, είναι και ε, η αρμόδια αρχή, η χώρα μέλος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι υπάρχει ένας διαχωρισμός, έτσι ώστε, λέει δηλαδή, σωστός διαχωρισμός μεταξύ συγκρουόμενων λειτουργιών. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ του ανάδοχου του σχεδίου και της αρχής που θα πρέπει να παράσχει τις πληροφορίες. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των επιπτώσεων. Η χώρα μέλος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Αυτό λέει και αυτό ακριβώς θα πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. Όχι μόνο αυτό. Θα πρέπει η εφαρμογή να γίνει σε επίπεδο αρχών. Ελπίζω να υπήρξα σαφή στην απάντησή μου. Η δεύτερη ερώτηση από το την βουλευτή από την Ιταλία. Ε, έχασα ένα μέρος της ερώτησής σας γιατί δεν πρόλαβα να βάλω το ακουστικά μου. Νομίζω ότι η ερώτησή σας ήταν παρεμφερής, αφορούσε διάφορα επίπεδα διακυβέρνηση και πού λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ε, μπορώ να σα παρακαλέσω να την επαναλάβετε. Η πρώτη μου ερώτηση αφορούσε τον ορισμό ενός ε, μιας πιο ολοκληρωμένη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου θα συμπεριλαμβάνεται και μια πιο μακρόπτωη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Γιατί πολλές φορές ε, δεν μπορεί να υπάρξει και μία παράλληλη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Και το δεύτερο μέρος της ερώτησης αφορά τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, πόσο εμπλέκονται σύμφωνα με την οδηγία στον έλεγχο και την παρακολούθηση του ε, έργου Νομίζω σημαντικό στόχος της οδηγίας είναι να εξασφαλίσει τον συνυπολογισμό θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον και να προωθήσει την βιώσιμη ανάπτυξη. Αν ληφθούν υπόψη κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα, θα πρέπει να θεωρηθούν ως θέματα που αφορούν άμεσα το περιβάλλον. Ο στόχος της οδηγίας είναι η περιβαλλοντική προστασία. Στο άρθρο 5 και στο άρθρο 8α είναι σαφές ε, τι θα πρέπει να είναι η απόφαση για τη χορήγηση άδειας οικοδόμησης. Δηλαδή θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα αν μπορεί να εφαρμοστεί ένα σχέδιο ή όχι. Θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι διάφοροι παράγοντες που αφορούν το περιβάλλον. Θα πρέπει να γίνει μία αξιολόγηση. Θα πρέπει να παρατεθούν οι λόγοι για τους οποίους ελήφθη μία απόφαση, πληροφορίες για μέτρα παρακολούθησης. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν έτσι ώστε όλοι να καταλάβουν. Όλοι να έχουν πληροφορίες για ποιο λόγο θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση. Νομίζω, ε, μάλλον ήθελα να σας πω ότι όλο το άρθρο 8α είναι καινούριο Εάν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο και εφαρμοστεί, θα μπορέσει να παράσχει εγγύησης για μία οδηγία που θα προωθεί την βιώσιμη ανάπτυξη και έτσι ώστε θέματα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά θα ληφθούν εξίσου υπόψη. Σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση, είναι αλήθεια ότι τα περισσότερα προγράμματα αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο. Συνεπώς η αρμόδια αρχή που θα πρέπει να αποφασίσει θα πρέπει να είναι τοπική. Μερικές φορές αυτό δημιουργεί θέματα ή οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων. Αλλά το γεγονός ότι η οδηγία απαιτεί την υποβολή ε, περισσότερων πληροφοριών στο κοινό, τη δημοσιοποίηση περισσότερων πληροφοριών για το κοινό πλην ληφθεί η απόφαση και οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να ανέβουν στην ιστοσελίδα των αρμόδιων αρχών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο εξασφαλίσει το ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη πληροφόρηση. Παράλληλα όμως θα πρέπει να δοθούν πληροφορίες, στοιχεία, ποιοτικά και ποσοτικά στην Επιτροπή κάθε έξι χρόνια με βάση μια έκθεση. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος μέλος θα πρέπει να δημιουργήσει ένα σύστημα για τη συγκέντρωση πληροφοριών από το τοπικό στο εθνικό επίπεδο προκειμένου να διαβιβαστούν στην Επιτροπή. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη το πώς θα συγκεντρώσουν τις πληροφορίες αυτές τα κράτη-μέλη από το τοπικό στο εθνικό επίπεδο δεν αναφέρεται στην οδηγία. Το γεγονός όμως ότι οι χώρες μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν αυτό το σύστημα επικοινωνίας μεταξύ του τοπικού και του εθνικού επίπεδου δίχως άλλο θα βελτιώσει την διακυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο γιατί θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Το σημαντικό είναι το να συμβεί, έτσι ώστε μετά από έξι χρόνια να μην βρεθούμε μπροστά σε μια κατάσταση που τα κράτη-μέλη θα πούν ότι δεν έχουμε πληροφορίες γιατί δεν μπορούν να συγκεντρωθούν πληροφορίες από τοπικό επίπεδο. Και αυτό έχει σχέση και με την οδηγία περιβαλλοντικής υπευθυνότητας εμείς έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα προκειμένου να συγκεντρώσουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα για την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ελέγχουν την εφαρμογή της νομοθεσίας που έχει εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ωραία. Ευχαριστώ. Ε, δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Από ό,τι βλέπω, Έχω λοιπόν τη χαρά να σας παρουσιάσω τον επόμενο ομιλητή. Είναι η κυρία Σάρα Ντρέικ. Είναι από τη νομική σχολή του Κάρντιφ και ο τίτλος από την Ουαλία, το τίτλος παρουσίασής της είναι εφαρμογή του κανονισμού του 2004 για τα δικαιώματα των επιβατών εναερίων μεταφορών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ονομάζομαι Δ. Σάρα Ντρέικ και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας μιλήσω για, για την οδηγία για τα δικαιώματα επιβατών αερομεταφορών. Θα επικεντρωθώ κυρίως στη μεταφορά της Εθνικό και την εφαρμογή. Η παρουσίασή μου χωρίζεται σε δύο τρίνα. Τα καταρχήν θα σας ενημερώσω για το ε, πεδίο εφαρμογή ε, και το έβρος του κανονισμού εφαρμογή και αδυναμίες, καθώς και την παρούσα κατάσταση. Και στο δεύτερο τμήμα θα επικεντρωθώ σε τέσσερις τομείς. Ε, θα μπορούσαμε να προτείνουμε κάποιες βελτιώσεις και θα παρουσιάσω και συστάσεις προς τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχήν να πω ότι κατά την αρχή της παρουσίασης ενώ η ανάλυση των περιπτώσεων στηρίζεται στα, πιο σύγχρονα διαθέσιμα στοιχεία, καθώ και κάποιες εκ των υστέρων του κανονισμού που έγιναν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, όλα αυτά υπάρχουν κάποια κενά στη συγκέντρωση των δεδομένων. Κάτι που καθιστά δύσκολη την ε, πλήρη εικόνα και την γενική επισκόπηση για την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ε-, ΕΟΧ. Ε, και θα σα μιλήσω και για τα στοιχεία που έχει η Επιτροπή Αναφορών σε ό,τι αφορά τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι πολίτε κατά την απόλαυση των δικαιωμάτων του. Ε, το σύστημα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία δικαιωμάτων αερομεταφορών είναι από τα πιο εκτενή στον κόσμο και δίνει άμεσα εφαρμοστέα δικαιώματα στους ε, επιβάτες που μπορούν να επικαλεστούν σε εθνικά δικαστήρια σε περίπτωση παραβίασης. Και η σχετική νομοθεσία είναι από τι εμβληματικέ πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με τον κανονισμό για τα τέλη περιαγωγή και πρόσφατα το Γενικό Κανονισμό Προστασία των Δεδομένων. Ο στόχο ε, του κανονισμού για τα δικαιώματα επιβατών αερομεταφορών είναι να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασία καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χορηγώντα δικαίωμα αρρωγή και αποζημίωση στου επιβάτε αερομεταφορών όταν ε, το ταξίδι του διαταράσσεται από άρνηση επιβίβαση, ε, ακούσια αναβάθμιση υποβάθμιση, καθυστέρηση ή ακύρωση. Επίση, οι αεροπορικέ εταιρείε οφείλουν να ενημερώνουν του πολίτε τους, τους επιβάτες για τα δικαιώματά τους. Και επίσης μπορούν ε, να αποκλείσουν την υποχρέωση αποζημίωσης όταν η διαταραχή του ταξιδίου οφείλεται σε εξαιρετικές έκτακτες περιστάσεις. Δηλαδή, αν δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί, ακόμη και αν είχαν λυθεί όλα τα λογικά μέτρα από τις αεροπορικές εταιρείε. Παρ' όλα αυτά, από την αρχή ε, δεν έγινε συμμόρφωση με τον κανονισμό. Είχαμε φυστέκες εκρήξεις, χιονοθύελες, αερο, ε, και ελλείψεις στον έλεγχο και κυκλοφορία. Γενικώ οι, οι επιβάτες προσπαθούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, αλλά δεν είναι εύκολο να λάβουν αποζημίωση ή να τα αποκαταστήσουν. Και μάλιστα παρεμποδίζονται από μη συνεργάσιμε και φιλόδικε αεροπορικέ εταιρείε, από αδύναμες δημόσιες αρχές εφαρμογής και κακώς ενημερωμένα δικαστήρια. Ε, επίσης, οι επιβάτες ε, στρέφονται προς ε, εταιρείε διαχείρισης τέτοιων ε, αξιώσεων, γιατί είναι αδύνατο μόνο τους να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Επίσης, γίνεται μια αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων εφαρμογής του κανονισμού στους εθνικούς φορείς επιλογής, επιβολής. και τα κράτη-μέλη θα πρέπει, οφείλουν να θεσπίσουν κάποιες κυρώσει που θα είναι αποτελεσματικέ, αποτρεπτικέ και αναλογικέ. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει σημαντικέ προσπάθειε να βελτιώσει το βαθμό εφαρμογή και να παροτρύνει τι ευρωπαϊ... ευρωπαϊκέ εταιρείε, ε, τι αεροπορικέ εταιρείε να συμμορφωθούν. Επίση υπάρχει και η πιθανότητα εναλλακτική επίλυση διαφορών. Η αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου ενημέρωσε το 75% των ε, καταγγελιών που, που έγιναν ε, στα πλαίσια του, της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών δικαίωσα τους επιβάτες. Βέβαια, η πρόσφατη αξιολόγηση και του ελεκτικού συνεδρίου της 8 η Νοεμβρίου του 2018 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δικαιωμάτων των Επιβατών είναι καλά σχεδιασμένο, αλλά ε, θα απαιτούν σημαντικές προσπάθειες για να μπορέσουν να υποφεληθούν από το σύστημα αυτό οι επιβάτες. Και ε, στις ε, έρευνες που έγιναν το 2015 με 2017 φάνηκε μεγάλο αριθμό καταγγελιών που γίνονται στου αρμόδιου φορείς επιβολή. Το 2017 αναφέρθηκαν πολλές περιπτώσεις συμμόρφωσης. Ε, βέβαια έγινε μια προσπάθεια το 2013 για αναδιατύπωση του κανονισμού προκειμένου να αντιμετωπιστούν κάποιε αδυναμίες ε, και να αντιμετωπιστούν οι λόγοι τη μη συμμόρφωση. Εκεί ε, ανα, ανακαλύφθηκε ότι δεν υπάρχει ένα ομοιόμορφο και αποφασιστικό σύστημα επιβολής ε, εφαρμογής στα κράτη-μέλη ε, και υπάρχει ένα μεγάλο κανονιστικό άχθος προς τις ε, αεροπορικές εταιρείες που είναι αντικίνητρο για την συμμόρφωση. Επίσης, κόλλησαν κάποιες αποφάσεις στο Συμβούλιο λόγω της διαμάχης μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ισπανία. Βέβαια, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου το 2019 ίσω ξεμπλοκάρει την νομοθετική διαδικασία. Και μάλιστα, ίσω αυτή είναι επίκαιρη εξέλιξη ε, μια και το σύστημα ε, ε, αντιμετωπίζει προβλήματα. Και μάλιστα το 2018 είχαμε σημαντικές καθυστερήσεις λόγω κακοκαιρίας, απεργιών και λήψεων στις, στον έλεγχο αέριο κυκλοφορίας. Κάτι που το κόστος για τις αεροπορικές εταιρείες παρόλο που δεν έφταιγαν. Και μάλιστα τον Ιούλιο του 2018 οι τέσσερι μεγαλύτερε αεροπορικέ εταιρείε έκαναν μια κοινή καταγγελία προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέγοντα το κλείσιμο του ενέργειου χώρου τη Γαλλία παρεμπόδισε το δικαίωμα ελεύθερη κυκλοφορία. Και μάλιστα με πρόβλεψη μεγέθυνση του κλάδου 5% κάθε χρόνο μέχρι το 2030 και με σημαντικέ ανησυχίε για την έλλειψη ικανότητα τη αγορά, η πλήρης απόλαυση των δικαιωμάτων των επιβατών αερομεταφορών φαίνεται ότι υπόκειται σε όλο και μεγαλύτερο κίνδυνο. Στο δεύτερο τμήμα τη παρουσίασή μου θα εντοπίσω πέντε τομεί που χρήζουν βελτίωσης και θα κάνω συστάσει και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, και από τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Ελήψη νομοθετικής αναθεώρησης, οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013 ε, στην προσπάθειά της ε, για τη διόρθωση, δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Έχουμε πρόβλημα με τη συνειδητοποίηση εκ μέρους των επιβατών και τη γνώση τους, ασφάλεια δικαίου, ε, εθνικά καθεστώτα επιβολής, ε, μονομένη επιβολή και αποκατάσταση και κανονιστικό βάρος προς αερομεταφορές. Ό,τι αφορά το πρώτο θέμα, συνειδητοποίηση και γνώση των επιβατών. Σίγουρα θα πρέπει οι επιβάτες να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Η διαμεσολαβήτρια κυρία Οράιλη επισήμανε τη σημασία που έχει η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα δικαιώματά τους. Το, το είπε νωρίτερα στην ομιλία της και είπε πόσο σημαντικό είναι αυτό εν ώψη και των ευρωεκλογών που θα γίνουν το Μάιο του 2019. Ο κανονισμός απαιτεί από τις αεροπορικές εταιρείες να ενημερώσουν τους επιβάτες για τα δικαιώματά τους. Πρόσφατη όμως έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου ε, διαπιστώνει ότι είναι πολύ χαμηλή αυτή η ευαισθητοποίηση των πολιτών. Μόνο 39% όσων έχουν ερωτηθεί από το ελεκτικό συνέδριο δηλώνουν ότι γνωρίζουν τα δικαιώματά του. Επίση, η έρευνα του Ελεκτικού Συνεδρίου αποκάλυψε ότι δεν είναι πάντα σωστή γνώση που έχουν οι επιβάτες για τα δικαιώματά του. Προτείνω λοιπόν τα Εθνικά Κοινοβούλια να φροντίσουν ότι, ώστε οι εθνικοί φορεί επιβολή να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση υποχρέωση παροχή πληροφορία και να λάβουν κάποια βήματα για να προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, τη συνειδητοποίηση εκ μέρου των επιβατών. Το Ελεκτικό Συνέδριο αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε πολλέ δράσει για να προωθήσει αυτή την ευαισθητοποίηση. Διαπιστώνει όμω ότι κάποιε ε, κατευθυντήριε γραμμέ στο διαδίκτυο δεν ε, εξηγούν με σαφήνεια πόσο, πώς πρέπει να αντιδρούν σε περίπτωση διαταραχή του ταξιδιού του οι επιβάτε. Επίση, προτείνει 10 συστάσεις ε, το ελεκτικό συνέδριο προ του Ταξιδιώτε σε περίπτωση διαταραχή του ταξιδιού. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια δικαίου, σίγουρα έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα, γιατί υπάρχουν κάποιες σαφέ ζώνε στον κανονισμό. Δηλαδή διατάξεις που είτε τη χάνουν συσταλτικής ή διασταλτικής ερμηνείας, για παράδειγμα η διασταλτικης ερμηνεια για παραδειγμα η εννοια των έκτακτων περιστάσεων και σχετικές εξαιρεσει. Και παρά τις πολύκροτες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εξακολουθεί να υπάρχει μια έλλειψη ασφάλειας δικαίου με μεγάλο αριθμό διαφορών μεταξύ αεροπορικών εταιριών και επιβατών. Επίσης ο κανονισμός είναι ιδιαίτερα περίπλοκος και μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για τους ενδιαφερόμενους να εντοπίσουν σωστά τα δικαιώματά τους. Για να βελτιωθεί λοιπόν η ασφάλεια δικαίου, οι αρμόδιοι εθνικοί φορεί επιβολή θα πρέπει να εξασφαλίζουν μια ενεργό συμμετοχή του στην ενημέρωση των επιβατών για τα δικαιώματά του, στι δυνατότητε που έχουν επανόρθωση, αποκατάσταση σε περίπτωση διαταρχή του ταξιδιού. Όταν τον Ιούλιο του 2018 η αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου για την πολιτική αεροπορία εξέδωσε κοινοθέντα τύπου με διευκρίνηση των δικαιωμάτων των επιβατών υπό το ενωσιακό δίκαιο μετά τι απεργίε τη Ryanair. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό και θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει με τις κατευθυντήριες γραμμές της ε, να εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου. Επίσης, χρειάζεται κατάλληλη κατάρτιση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του κανονισμού στο εθνικό δίκαιο για να δημιουργηθούν ικανότητες ε, που θα μπορούσαν να διευκολυνθούν από τα Εθνικά Κοινοβούλια και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Τρίτο στοιχείο. Τα εθνικά συστήματα για την επιβόλη του κανονισμού. Σημαντικές αδυναμίες εντοπίζονται εκεί σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του κανονισμού. Μάλιστα, ο κανονισμός... Ε, δίνει υπερβολική διακριτική ευχέρεια στα κράτη-μέλη, κάτι που οδήγησε σε διαφορετικά επίπεδα εφαρμογής. Ακόμη πιο σημαντικό όμως, πολλά εθνικά καθεστώτα επιβολής παρά είναι αδύναμα για να αποτρέψουν τη μη συμμόρφωση στις αεροπορικές εταιρείες. Βασικές αδυναμίες είναι ανεπαρκής πόροι, έλλειψη τεχνικής και επιχειρησικής εμπειρογνωμοσύνης για να ε, εξεταστεί η εγκυρότητα της εξαίρεσης των εκτακτών περιστάσεων. Δεν είναι αρκετά υψηλέ οι κυρώσεις για να είναι αποτρεπτικές και μάλιστα λιγότερο από 1000 ευρώ είναι η μέσος, ο μέσος όρος του προστήμου σε τέτοιες περιπτώσεις όπως λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, δεν είναι αρκετά προορατικές οι εθνικές οργανώσεις. Ε, και το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε ότι τα εθνικά, οι εθνικοί φορείς ε, δεν τιμωρούσαν τη μη συμμόρφωση συστηματικά, παρά μόνο 1 με 2% των περιπτώσεων ε, τιμωρούνταν. Επίσης, τα κατόφλια μερικές φορές δεν τηρούνται για την επιβολή ε, κυρώσεων, γιατί μερικές φορές πρέπει να ακολουθεί ποινική διαδικασία και όχι απλώς διοικητική διαδικασία. Σε κάποιες χώρες οι εθνικοί φορείς επιβολής δεν έχουν την ικανότητα να προτείνουν με, μεμονωμένα μέτρα αποκατάστασης και υπάρχουν και νομικές ή και πρακτικές ε, δυναμίες προκειμένου να εφαρμοστούν οι κυρώσεις που θεσπίζονται στα κράτη-μέλη ή να ε, εισπραχθούν τα πρόστιμα από αερομεταφορές που βρίσκονται σε άλλα κράτη-μέλη. Επίσης, η ερμηνεία του κανονισμού από τους, εθνι... από τους εθνικούς φορείς επιβολής, κυρίως για την έννοια των... της εξαίρεσης των έκτακτων περιστάσεων, είναι πολύ διαφορετική. Και το επίπεδο των ερευνών επίσης είναι διαφορετικό. Ίσως λοιπόν αυτό είναι ένας ε, τομέας στον οποίο τα Εθνικά Κοινοβούλια μπορούν να συνεισφέρουν και να βελτιώσουν την επιβολή σε εθνικό επίπεδο. Χρειάζεται λοιπόν ε, να υπάρχει ε, αποτρεπτική ικανότητα έτσι ώστε οι αεροπορικές εταιρείες να συμμορφωθούν, να είναι δηλαδή πιο δαπανηρό οικονομικά να παραβιάζουν την νομοθεσία από ότι να την ακολουθούν. Οι επιβάτες επίσης πρέπει να, ακολουθούν, να έχουν δυνατότητα προσφυγής σε ένδικα μέσα και να μην υπάρχει ατιμορρησία για τις αεροπορικές εταιρείες που παραβιάζουν. Χρειάζεται λοιπόν ε, νομοθεσία που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των αεροπορικών ε, επιβατών πρέπει να ξεκινήσουν με κάποιο, κάπως πιο μέτριες παρεμβάσεις που στόχο έχουν να αυξήσουν τη συμμόρφωση και έπειτα ε, να αυξάνονται οι ποινές, να γίνουν πιο τιμωρητικέ. Οι εθνικές αρχές επιβολής της Ολλανδίας μάλιστα πρότειναν μια κλιμακωτή αντιμετώπιση και αυτό βρίσκεται στο ενημερωτικό σημείωμα ε, υπό τον τίτλο «Πυραμίδα επιβολής» που σας δείχνει ακριβώς πόσο μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο σχέδιο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τι συστάσεις, τα εθνικά κοινοβούλια θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην ε, διασφάλιση ε, της ε, επιβολής τόσο της εθνικής πολιτικής όσο και του εθνικού πλαισίου, της επιβολής αλλά και της προσαρμογής τους έτσι ώστε να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν αυτόν, αυτήν την νομοθεσία που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες προκύπτουν. Μετά, η αποτελεσματική επιβολή προϋποθέτει οι επιβάτες να έχουν τη δυνατότητα προσφυγή σε ένδικα μέσα για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Και αυτός είναι ένας χώρος στον οποίο έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις, για παράδειγμα με την χρήση της εναλλακτικής διευθέτησης διαφορών, που επιτρέπει στους επιβάτες να ε, έχουν ε, πρόσβαση σε, ε, σε αποτελεσματική αρρωγή. Χρειάζεται όμως καθοδήγηση για τις διαφορετικές επιλογές που έχουν οι επιβάτες, για τα ωφέλη και τα μειονεκτήματα και επίση την προώθηση της εναλλακτική διευθέτησης διαφορών, μια που είναι γρήγορη, αποτελεσματική και οικονομική. Το 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε δυνατή τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πάνελ αρμόδιων φορέων για τις αεροπορικές μεταφορές ως ένα βήμα ανταλλαγής απόψεων και των πρακτικών. Αυτό δίνει την δυνατότητα διευκόλυνσης ε, της συλλογής στατιστικών ε, στοιχείων ε, σχετικά με την επιβολή του κανονισμού 261 στα, κράτη, στα διάφορα κρατημέλη. Ένα αποτρεπτικό παράγοντα προσφυγή στο δικαστήριο είναι ότι ε, αυτό είναι χρονοβόρο και με μεγάλο κόστος. Ε, τα συλλογικά ένδικα μέσα είναι στο πλαίσιο μια νέα συμφωνία για του καταναλωτέ που θα του ε, δίνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τι παραβιάσεις του κανονισμού 261. Αυτό είναι κάτι που έχει βρει πολύ μεγάλη αντίσταση από τι αεροπορικέ εταιρείε, αλλά έχει στηριχθεί πολύ και από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου και από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ε, υπάρχουν αρκετέ ε, συζητήσει ε, για το αν η αποζημίωση θα πρέπει να γίνεται αυτόματα. Τον Ιανουάριο του 2018 η Ράινερ δήλωσε ότι διερευνά και εξετάζει το ενδεχόμενο αυτό, αν και θα επιφέρει ίσω πρόσθετο κόστο και διοικητικό άχθο για τι αεροπορικέ εταιρείε. Βέβαια, το δικαστήριο έχει μπορεί να προβλέψει υποχρεωτική αποζημίωση. Ενώσεις καταναλωτών έχουν πρόσφατα ξεκινήσει εκστρατεία έτσι ώστε να εγκριθεί αυτή η νομοθεσία και έχουν συλλέξει εκατοντάδες χιλιάδες υπογραφές. Περνάμε τώρα στον τελευταίο τομέα που προκαλεί ανησυχίες, είναι η διαχείριση του, ε, ρυθμιστικού φόρτου από τι αεροπορικέ εταιρείε. Ε, υπάρχει πίεση συμμόρφωση προ τον κανονισμό σε, περίπτωση, σε περιπτώσεις που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους. Για παράδειγμα, η παροχή φροντίδας και σε που ε, σε επιβάτες ε, μετά από ακυρώσεις πτήσεων λόγω, για λόγους ανωτέρας βίας. Αυτό έχει πολλές διοικητικές και οικονομικές επιπτώσεις για τις αεροπορικές εταιρείε. Τα εθνικά κοινοβούλια όμως θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει η δυνατότητα αντίδραση στον χώρο των αερομεταφορών έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν λήψεις του εργατικού δυναμικού, απεργίες ή διάφορα άλλα ε, φαινόμενα που εμποδίζουν τις αεροπορικές μεταφορές. Όμως ε, αυτό είναι σχεδόν αδύνατον. Συμπληρω... Συμπερισματικά λοιπόν Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που υπονομεύουν το υψηλό επίπεδο προστασίας καταναλωτών που προσπαθεί να ε, δώσει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στου επιβάτε ε, των αερομεταφορών. Η επιβολή του κανονισμού 261 είναι αποκεντρωμένη, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ε, διασφαλιστεί ότι τα κράτη-μέλη θα, εφαρμόζουν, θα εφαρμόσουν σωστά τον κανονισμό και θα υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι γι' αυτό. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα επίση ενδεχομένω έχουν την ευκαιρία να επανεξετάσουν το νομικό πλαίσιο του κανονισμού 261 και να στηρίξουν τι συστάσει έτσι ώστε να ε, διευκρινιστούν τα δικαιώματα και υποχρεώσει, να ε, εξισορροπηθεί ο ο ρυθμιστικός ε, φόρτος και να βελτιωθεί η επιβολή. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα πλαίσιο για, ε, έτσι ώστε να μπορούν να ε, προσφεύγουν μεμονωμένα οι επιβάτες και να υπάρχουν κίνητρα για τις αεροπορικές εταιρείες να συμμορφώνονται με τον κανονισμό. Όμως ο ρόλος της μεμονωμένης προσφυγής ένδικα μέσα είναι να συμπληρώνει την εθνική επιβολή και όχι να την υποκαθιστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, ε, ε, ακούσαμε και την ε, τελευταία παρουσίαση σήμερα το πρωί και θα ήθελα τώρα να ανοίξω τη συζήτηση, να δώσω το λόγο σε εσά για ερωτήσει ή σχόλια. Ποιο θα ήθελε λοιπόν το λόγο για ερώτηση ή σχόλιο. Κανείς. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Νομίζω λοιπόν πως τώρα έφτασε η ώρα να κλείσουμε το πρώτο πάνελ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ιδιαίτερα τους προσκεκλημένους. Ευχαριστώ πολύ και όλους τους παρευρισκόμενους. Έχω πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά νέα. Θα ήθελα λοιπόν να προσκαλέσω όλους εσάς όλους τους παρευρισκόμενους ε, σε ένα γεύμα το οποίο παραθέτει η Ευρωπαϊκή Διαμεσολαβήτρια, το οποίο θα γίνει στην Μπρασερή, στο εστιατόριο του τρίτου ορόφου, εδώ σε αυτό το κτίριο. Όποιος ε, δεν γνωρίζει υπάρχουν μέλη της Επιτροπής Αναφορών ε, που είναι πρόθυμα να σας βοηθήσουν. Στο εστιατόριο λοιπόν, στον τρίτο όροφο αυτού του κτίριου, θα παρατεθεί γεύμα από τις 2... Όχι, όχι, όχι, όχι, από τις 2, με συγχωρείτε, σε 35 λεπτά, στις 12.30, στον τρίτο όροφο του στο εστιατόριο. Θα συνεχίσουμε στις 2.30, εδώ σε αυτή την αίθουσα. Γι' αυτό λοιπόν σας εύχομαι καλή όρεξη και θα τα πούμε στις 2.30. Εδώ. Σας ευχαριστώ.